Good morning everybody. I think we are just... Καλημέρα σας. Είμαστε Pani marszałek, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι. Θα συμπροεδρεύσω στη συζήτηση για την ευρωπαϊκή πολιτική ισότητα ε, των φύλων και των δημογραφικών αλλαγών. Ξεκινώντας θέλω να κάνω μια παρατήρηση. θα πρέπει να ορίσουμε την έννοια της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών σήμερα δεν είναι μονόδρομος. Όχι μόνο. Οι νέοι θα πρέπει να είναι αλληλέγγυοι έναντι των ηλικιωμένων, αλλά και οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να είναι αλληλέγγυοι έναντι των νέων. η γενεά μεταξύ των 30-40 ετών, η γενεά Χ, όπως ορίζεται, είναι, βρίσκεται σήμερα σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Πρόκειται για μία γενεά η οποία θα πρέπει να υλοποιήσει τις φιλοδοξίες της, θα πρέπει να κερδίσει χρήματα, αλλά θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην επιχορήγηση των ταμείων για την καταβολή των συντάξεων ε, των παππούδων, ε, των γονέων κλπ. Και να προβλέψει φυσικά και τον, το μέλλον των παιδιών της. Είναι μια γενεά η οποία δεν εργάζεται πια για τον εαυτό της. Είναι φανερό ότι η ευρωπαϊκή πολιτική, οικονομική και κοινωνική αντιμετωπίζει πρόβλημα. Για να βελτιώσουμε τη δημογραφική κατάσταση είναι θεμελιώδες όχι μόνο να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής των ηλικιωμένων αλλά να αυξήσουμε και την γεννητικότητα. Η δημογραφική ανανέωση είναι η μόνη στρατηγική μακροπρόθεσμα που θα μπορέσει να μας βοηθήσει σε πολιτικό επίπεδο και πρέπει να την προωθήσουμε. Όλες οι χώρες έχουν χαμηλά επίπεδα γεννητικότητας. Ακούσαμε να... Στο πρώτο και στο δεύτερο πάνελ ακούσαμε για την Αγγλία και την υπογεννητικότητα. Τι να κάνουμε λοιπόν. Πώς μπορούμε εμείς ε, να διδαχθούμε από τις εμπειρίες των άλλων χωρών. Οι μελέτες αποδεικνύουν ότι τη μεγαλύτερη γεννητικότητα την έχουμε στις χώρες εκείνες όπου υπάρχει ισότητα των φύλων, όπου καταμερίζονται, καταμερίζονται οι αρμοδιότητες στην οικογένεια. Και εκεί όπου υπάρχουν μέτρα στήριξης υπέρ των οικογενειών για το μεγάλωμα των παιδιών. Η δημογραφική πολιτική, η δημογραφική ανανέωση, η πολιτική για τις οικογένειες είναι μια πολύ δάπανη πολιτική. Για αυτό πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσο τα ευρωπαϊκά προγράμματα θα πρέπει να υποστηρίζουν τις πολιτικές των κρατών μελών και των περιφερειών για την υλοποίηση αυτών των πολιτικών. Πολλές φορές ε, λείπουν ε, τα, τα κονδύλια και δεν είναι καθόλου εύκολο. Στο πρώτο πάνελ ε, φάνηκε ότι η καλύτερη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε για τις δημογραφικές αλλαγές ε, είναι να οδηγήσουμε τους ηλικιωμένους να εργάζονται περισσότερο. Αλλά αυτό όμως άμα θα έχουμε και την κατάλληλη πολιτική για να απασχολήσουμε αυτούς τους ηλικιωμένους. Αδιαμφισβήτητα δεν πρόκειται εδώ μόνο για μια υπόθεση αγοράς εργασίας, πρέπει να έχουμε μια οριζόντια προσέγγιση τη λεγόμενη mixed policy. Θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την καινοτομία, την εκπαίδευση, την πολιτική στον τομέα της υγείας. Η αγορά εργασια σήμερα είναι εντελώς διαφορετική από πριν από ότι πριν από μία δεκαετία αλλά και πριν από μερικά χρόνια ε, τα πράγματα ήταν διαφορετικά αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα ο κόσμος και οι νέες γενιές αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα στην ανταγωνιστικότητα, διότι αυτοί οι πολλοί νέοι ανταγωνίζονται για μια θέση εργασίας με ανθρώπους πολύ πιο ηλικιωμένους. Πρόκειται για μια πρόκληση το θέμα της απασχόλησης των ηλικιωμένων χωρίς στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης για την τρίτη ηλικία. Δεν θα είμαστε σε θέση να καταφέρουμε οι ηλικιωμένοι να εργάζονται παραπάνω. Η φλέξη ασφάλεια λειτουργήσε για την απασχόληση των γυναικών και των νέων. Κυρίως για τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίες θα πρέπει να γυροκομίσουν γονείς, συγγενείς κλπ. Η αύξηση όμως της ανεργίας έπληξε κυρίως τους ηλικιωμένους και τις γυναίκες. Και αρχίζουμε και απομακρυνόμαστε από τους προκαθορισμένους στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020. Πρέπει να κάνουμε κάτι ώστε οι ηλικιωμένοι και κυρίως οι γυναίκες να μην χάσουν τα ευεργετήματα τα οποία έχουν ε, από το σύστημα προνοίας. Και υπάρχει και ένα άλλο εμπόδιο το οποίο θα πρέπει να ξεπεράσουμε. Είναι η ελάχιστη διάθεση που δείχνουν οι εργοδότες να προσλάβουν ηλικιωμένους. Πρόσφατα ολοκληρώσαμε μια μελέτη στην Πολωνία και διαπιστώσαμε ότι ακόμη και οι μεγάλες πολυεθνικές έχουν πρόβλημα να καταλάβουν ότι στις πολιτικές τους απασχόλησης στο θέμα της διαχείρισης των κατηγοριών ηλικίας είναι θεμελιώδες. Η Πολωνία και η Ιταλία έχουν εμπειρία επίσης στην απασχόληση των ανέργων μακριάς διαρκείας. Και μεταξύ αυτών έχουμε ηλικιωμένους και γυναίκες. Έχουμε θετικές εμπειρίες στην εφαρμογή της αρχής της, κοινωνική, της λεγόμενης κοινωνικής απασχόλησης. Υπάρχουν κέντρα κοινωνικής ενσωμάτωσης, κοινωνικής ένταξης. Θα έπρεπε ίσως σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ευνοήσουμε αυτόν τον νέο τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Στην Πολωνία έχουμε το πρόγραμμα 50 και πάνω για τους ηλικιωμένους. Άρχισε να εφαρμόζεται αυτό το πρόγραμμα, αλλά λόγω της κρίσης δεν θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους που είχαμε θέσει. Χρειαζόμαστε νέα κίνητρα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται επίσης μέσα για να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες για την ολοκλήρωση αυτών των κοινωνικών πολιτικών. Το πρώτο μέσο είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ακούσαμε διάφορα σχέδια σχετικά, ούτως ώστε οι δαπάνες για τις πολιτικές σύνοχης να περικοπούν. Φοβούμε ότι αυτές οι περικοπές θα ισχύσουν και για το κοινωνικό ταμείο. Δεν θα πρέπει όμως να συμφωνήσουμε με αυτή την περικοπή των πόρων του κοινωνικού ταμείου. Κυρίες και κύριοι, αν εμείς σήμερα δεν παρέμβουμε στην αγορά εργασίας, αν δεν ανταποκριθούμε στις δημογραφικές προκλήσεις, το κόστος αυτής της αμέλειας θα είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο στο μέλλον. από ότι τα πρόσκαιρα πλέον εκτήματα περικοπών. Θα πρέπει να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των πρωτοβουλειών μας και να επικεντρωθούμε γύρω από συγκεκριμένες προτεραιότητες. Υπάρχουν επίσης τα θέματα συντονισμού. Ορισμένοι αστευόμενοι λένε ότι πρόκειται απλά και μόνο για μια στατιστική μεθοδολογία, ευρωπαϊκή στατιστική μεθοδολογία. Για να μην μείνει όμως έτσι το πράγμα στάσιμο θα πρέπει να προωθήσουμε, να ενισχύσουμε όλους αυτούς που θέλουν να πετύχουν αυτούς τους στόχους. Οι ανάγκες των ηλικιωμένων διαφέρουν. Ε, πρόκειται για μια, για, ηλικία που ξεκινάει από τα 50 και πάει στα 90 ε, με διαφορετικές υποκατηγορίες και ανάγκες στο εσωτερικό της. Οι υποδομές για μια μακροπρόθεσμη βοήθεια, επικουρία των ατόμων με ειδικέ ανάγκες στοιχίζει πολύ. Ορισμένοι λένε ότι υποστηρίζοντας τις οικογένειες θα μειώσουμε αυτόματα τις ανάγκες για τις φροντίδες των ηλικιωμένων. Όχι, δεν ενισχύει αυτό. Πρέπει να βοηθήσουμε τα κράτη να αναπτύξουν αυτού του είδους τις υπηρεσίες, να θεσμοθετήσουν αυτού του είδους τις ε, υπηρεσίες, διότι στο μέλλον θα υπάρχει πάντα πολύ μεγαλύτερη ζήτηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν θα πρέπει να περιορίζεται στη χρηματοδότηση μόνο των μικρών σχεδίων. Θα πρέπει να υπάρχουν κονδύλια και για την ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών. ένα καλό λειτουργικό σύστημα για τις φροντίδες μακράς διαρκείας, αν είναι καλά οργανωμένο, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα νέο οικονομικό, ισχυρό οικονομικό τομέα. Στην Πολωνία, σε αυτόν τον τομέα δημιουργούνται πολλές νέες επιχειρήσεις. Αν εμείς θέλουμε να μειώσουμε μελλοντικό κόστος σε αυτόν τον χώρο, θα πρέπει να στοιχηματίσουμε στην ανάπτυξη αυτής της αγοράς. Πρέπει αυτή... Αυτός ο κλάδος μπορεί να δημιουργήσει τεράστιες, τεράστιο αριθμό θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέσεις εργασίας που μπορούν κάλλιστα να καλυφθούν από γυναίκες κοντά στην ηλικία σύνταξης. Μειώνει επίσης τις δαπάνες στον τομέα της υγείας. Οι ηλικιωμένοι έχουν μια τεράστια δυναμική μέσα τους. Το που πρέπει να κάνουμε είναι να δραχθούμε τις ευκαιρίες και να χρησιμοποιήσουμε την θετική ενέργεια αυτού του κύματος, αυτής της ομάδας ανθρώπων που βλέπουμε σε αυτή τη δημογραφική αλλαγή, δηλαδή των υπερηλίκων, των ηλικιωμένων. Και είναι δυνατόν κύριε και κύριοι και μπορεί να ωφελήσει και να είναι χρήσιμο αυτό για να υλοποιηθεί η ανάπτυξη, να επιτευχθεί η ανάπτυξη. Ένα παράδειγμα θα είναι του χρόνου, 2012 για τις δραστηριότητες των υπερηλίκων ηλικιωμένων στην Ευρώπη. Εμείς στην Πολωνία θέλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε στα διαφορετικά προγράμματα να κάνουμε ό,τι γίνεται για να τονίσουμε ιδιαίτερα την κατάρτιση, παιδεία, εκπαίδευση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα έχουμε τα πανεπιστήμια της τρίτης ηλικίας. Αυτές οι οργανώσεις, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, θα μπορέσουν να δράσουν και θα εργαστούν και θα συνεισφέρουν ιδιαίτερα στην Πολωνία. Έχουμε πολλά πανεπιστήμια, πολλά, που όχι μόνο με τους φοιτητές τους ε, υλοποιούν δράσεις ε, για να προωθηθεί ακόμα περισσότερο το δυναμικό των ε, ηλικιωμένων, αλλά έχουν και δραστηριότητες στον πολιτισμικό τομέα, στον τουριστικό τομέα, στον τομέα της ένταξης και ολοκλήρωσης. Δημιουργούν αυτόν τον δεσμό, αυτή την διασύνδεση μεταξύ των γενεών, ώστε να μπορούν να είναι αυτόνομοι και να δοθούν πορείες και κατευθύνσεις πώς μπορούν να γίνουν τα πράγματα καλύτερα, πώς μπορεί στην πολιτική να ενδυναμωθούν τα ίδια τα άτομα που είναι ηλικιωμένα. Διότι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες βλέπουμε το επίπεδο συμμετοχής των ηλικιωμένων όταν έρχεται η ώρα λήψης αποφάσεων βλέπουμε ότι είναι πολύ χαμηλό, υπερβολικά χαμηλό αυτό το επίπεδο. Και είναι σημαντικό και σε, αυτό το, σε αυτόν τον τομέα να βρούμε αυτές τις λύσεις για εκείνα τα ευρωπαϊκά κράτη όπου θα διασφαλίζεται ότι θα λαμβάνονται αποφάσεις για τους ηλικιωμένους με την δική τους την ίδια συμμετοχή των ηλικιωμένων. Και θα προαχθεί έτσι η ανάπτυξη των οργανώσεων ε, βοήθειας και στήριξης. Ε, και θα ολοκληρώσω για αυτό το θέμα και για αυτές τις πτυχές ε, που συσχετίζονται με, την δημογραφική, με τις δημογραφικές εξελίξεις της ε, όσον αφορά την απασχόληση και την ισότητα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρουσίασή σας και έχοντας ε, προβλέψει συζήτηση έχουμε μία ώρα και 15 λεπτά για τη συζήτηση συνολικά αυτών των τυχών. Κάποιος ήδη ζήτησε τον λόγο. Πρωτού ξεκινήσουμε τη συζήτηση, θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε έναν ειδικό κανόνα. Στην περίπτωση που θα έχουν ζητήσει αρκετοί τον λόγο να παρέμβουν, θα, έχετε, θα έχουμε δύο ευρωβουλευτές με δύο βουλευτέ από τα Εθνικά Κοινοβούλια, ένα ευρωβουλευτή και μετά θα συνεχίζουμε έτσι ένα λάξ. Έχετε όλοι μπλε κάρτε. Οπότε θεωρείτε ότι θα θέλατε να διατυπώσετε μια ερώτηση για μισό λεπτό με την μπλε κάρτα και αν η κάρτα μπορείτε να το κάνετε. Πρέπει για την προηγούμενη πάντα παρέμβαση να είναι αυτή η μπλε κάρτα. Σε σχέση με τον προλαλήσαντα, μια τέτοια ερώτηση μπορεί να έχει τη δυνατότητα να τύχει απάντηση. Λοιπόν, με αυτά μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ο πρώτος που ζήτησε να παρέμβει είναι ο κύριος Χέρμαν Ντεκρό από το Σώμα των Εκπροσώπων του Βελγίου. Oh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. καλώς ε, ήρθατε στις Βρυξέλλες. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στην πολιτική και στο κοινοβούλιο ήμουνα και υπουργό Παιδείας και υπουργό για τις συντάξεις και υπάρχουν αρκετά προβλήματα και ερωτήματα τα οποία μου τίθενται ακούγοντας την ε, τοποθέτηση του κυρίου Ογκοστά. Εμείς χρειαζόμαστε γυναίκες ε, στη δουλειά και νέους χρειαζόμαστε και ηλικιωμένους που εργάζονται περισσότερο χρόνο. Οι γυναίκες στη δουλειά πραγματικά Τις θαυμάζω πάρα πολύ, διότι όλες ασχολούνται σε διπλά επαγγέλματα. Στο επάγγελμα της μητέρας, ε, της συντρόφου, της, ε, της γυναίκας, ε, της γιαγιάς. Το θέμα της ύπαρξης παιδικών σταθμών είναι πάρα πολύ σημαντικό άμα θέλουμε να έχουμε γυναίκες στη δουλειά για τους νέους το πρόβλημα είναι πολύ πιο σοβαρό. Εμείς έχουμε ένα σωρό νέους που έρχονται στις χώρες μας και από χώρες μακρινές από την Ευρώπη. Και εγώ διαπίστωσα στο Υπουργείο Παιδείας ότι η κατάρτιση αυτών των νέων, ακόμη και αν όταν γίνονται Βέλγοι, και ή παίρνουν την υπηκότητα μία από τις χώρες μας είναι σύνθετη και δύσκολη. Τα σχολεία δεν είναι έτοιμα για την κατάρτιση αυτού του τύπου των νέων και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η ανεργία των νέων εκφράζεται μέσα από αυτούς τους μετανάστες πρώτης δεύτερης γενιάς οι οποίοι δεν μπόρεσαν να καταρτιστούν σωστά στα σχολεία. Το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό σοβαρό. Δεν μπορούμε εμεί μόνο να τους να ζητάμε από τους νέους να δουλέψουν. Εμείς θέλουμε να τους ζητήσουμε να δουλεύουν και παραπάνω χρόνο, διότι αυτό θα στοιχήσει λιγότερο στο σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων. Το μεγαλύτερο μέρος του των εισφορών μας ε, στις κοινωνικές ασφαλίσεις απορροφώνται τα τελευταία χρόνια της ζωής μας. Τώρα, αυτοί οι οποίοι ζουν περισσότερα χρόνια, ζουν πιο γέροι, στοιχίζουν ζουν πολύ πιο ακριβά. Και σε περίοδο ανταγωνισμού και κρίσης, Συγγνώμη που σας διακόπτω. Λυπούμε που σας διακόπτω, αλλά ξέχασα να αναφέρω κάτι πολύ σημαντικό. Τρία, όρια, τρία λεπτά είναι το όριο για την ερώτησή σας. Φυσικά οι πληροφορίες σας είναι πολύ επικοδομητικές, αλλά να προχωρήσουμε στην ερώτηση, γιατί και περιμένουν άλλοι να παρέμβουν. Ο μόνος ο τρόπος ε, να ε, μπορέσουμε να προχωρήσουμε είναι και με έκπληξη στρεφόμουν στο ε, γεγονός ότι δεν είχε υπάρξει αντίδραση. Λοιπόν, η ερώτησή μου είναι απλή. Τι κάνουμε όσον αφορά την παιδεία και την εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων, ιδιαίτερα εκείνων που έρχονται από το εξωτερικό. Τι κάνουμε και τι θα κάνουμε ώστε να καλυφθεί το, η διαφορά αμοιβών σε σχέση με την δυνατότητα να είναι πιο φθηνή στην απασχόληση όταν είναι 60-65 και να μην είναι πιο ακριβή σε σχέση με την ηλικιακή, το ηλικιακό τομέα των 35 άριδων. Πρέπει να αλλάξουν λοιπόν και οι αμοιβέ και το επίπεδο αυτό. Και το τελευταίο που θα ήθελα να αναφέρω είναι αυτό που είναι η τελευταία ερώτηση ε, το θέμα της ανάπτυξης, το θέμα της συμμετοχής. Ένα τέταρτο των εκλογέων είναι πάνω από 60 ετών. Αν σε ένα δημοκρατικό καθεστώς ε, σήμερα μια πλειοψηφία μπορέσει να ε, θεσπιστεί, πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι ένα τέταρτο των εκλογέων είναι πάνω από 60 ετών. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι οι ηλικιωμένοι έχουν και πρέπει να έχουν μια πιο ενισχυμένη θέση που θα ανήκει σε αυτούς σε ένα δημοκρατικό καθεστώς. Και θα πρέπει να σκεφτούμε, λέμε, ότι οι ηλικιωμένοι που έχουν καλή εκπαίδευση θα πρέπει ως εταίροι να χρησιμοποιηθούν για καλύτερη ανάπτυξη και των αναπτυσσόμενων χωρών μέσω της κατάρτισης και εκπαίδευσης. Θα μπορούσαμε στην Ευρώπη να σκεφτούμε ότι θα υπήρχαν ε, τέτοιοι άνθρωποι 60-65 ετών που θέλουν να συνεχίσουν να είναι δραστήριοι. Ευχαριστώ Πρόεδρε για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε τελικά, διότι θα γίνουμε τελικά η εσπερία που θα δύσει ο ήλιος και δεν θα ξανανατείλει. Σας ευχαριστώ. Τρία λεπτά είναι το όριο. Υπάρχουν τόσοι πολλοί που έχουν ζητήσει τον λόγο. Λοιπόν, εντάξει με την παρέμβασή σας και για την παρέμβαση και ερώτηση από πλευρά του Βελγίου. Τώρα, εσείς θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε παρακαλώ αυτή την ερώτηση. Έχετε τον λόγο κύριε. Ευχαριστώ. Είναι σαφές ότι δεν έχουμε μία ενιαία μοναδική απάντηση από πλευρά τη Ευρώπη σε αυτή την ερώτηση. Πώ δηλαδή θα προπαρασκευάσουμε και θα προετοιμάσουμε τα εκπαιδευτικά συστήματα για την κατάρτιση και εκπαίδευση και των μεταναστών αλλά και των ηλικιωμένων. Δεν υπάρχει βέβαια καμία αμφιβολία ότι αυτό θα έπρεπε να είναι ένα από του στόχου αυτή τη ανοιχτή μεθόδου συντονισμού μέσα στο πλαίσιο ακριβώς ανταλλαγής ε, ε, εμπειριών και πείρας. Θα πρέπει να επιλέξουμε τις καλύτερες, βέλτιστες λύσεις που σίγουρα έτσι θα μπορέσουν να εμπλουτίσουν, να εμπλουτίσουν τις χώρες μας. Όταν γίνεται λόγος για την υποστήριξη όσον αφορά την πρόσληψη ε, των ηλικιωμένων και τις μεγαλύτερες δαπάνες που συνεπάγεται ίσως αυτό στην αγορά εργασίας, θα ήθελα να πω τούτο. Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι δεν είμαι 100% σύμφωνος με αυτά τα οποία αναφέρθηκαν. Είναι βέβαια σαφές ότι πρέπει να δούμε μέχρι ποιου σημείου το να διατηρείται μια θέση απασχόλησης ή το να προετοιμάζεται μια τέτοια θέση απασχόλησης και όσον αφορά και τους όρους, όσον αφορά την κατάρτιση και την χρήση νέων τεχνολογιών, όλα αυτά είναι πολύ πιο δαπανηρά από την περίπτωση των νέων. Ίσως ναι, εντάξει, αλλά είναι μια παράμετρος που ίσως μπορεί να καταλήξει πιο μακροπρόθεσμα σε επιπτώσεις. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι είναι πολύ πιο πιστοί και εξάλλου οι αποδείξεις δείχνουν ότι ε, υπάρχει ε, λιγότερη απουσία από τους χώρους εργασίας ή λόγω ασθένειας ή λόγω απουσιών και όσον αφορά την κινητικότητα είναι πολύ περισσότερα στη διάθεση των εργοδοτών κτλ το δικό μας βίωμα, η πείρα στην Πολωνία δείχνει το εξής. Όταν υποστηρίζεται η πρόσληψη ηλικιωμένων, τότε μπορούμε να δρέψουμε, ε, να θερήσουμε καλούς καρπούς. Και βλέπουμε για το πρόγραμμα το οποίο αναφέρεται, για την ε, αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών για εκείνους που είναι πάνω από τα 50 χρόνια, είναι πλέον σαφές ε, και έχουμε και την απόδειξη για το τι συνέβη και λόγω της οικονομικής κρίσης έχουμε και πάλι τώρα ένα κύμα ηλικιωμένων εργαζομένων, πολλούς ηλικιωμένους εργαζόμενους χωρίς απασχόληση. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εκπαιδεύσουμε, να τους προετοιμάσουμε, να τους κατατήσουμε για να ξαναβρούν απασχόληση. Είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε μία μπλε κάρτα. Το όνομά σας παρακαλώ και θέστε την ερώτησή σας. Ευχαριστώ. Από την Βουλή, από ε, την συνέλευση της Πολωνίας, έχω αρκετούς ε, που έρχονται στα γραφεία μου ε, άνθρωποι, πολίτες με πάνω από 50 χρόνια όσον αφορά την ηλικία τους και θέλουν να δουν τι θα γίνει με αυτή την ανεργία. Όσον αφορά αυτά θα ήθελα να πω στον συνάδελφο ότι είναι εξαιρετική η πρόταση και θα έλεγα υπάρχει εδώ μεγάλο δυναμικό. Έχουμε και επαφή με εκείνους που απασχολούν τους ηλικιωμένους ε, σε σχέση με τις λιγότερες δαπάνες, μικρότερες κοινωνικές εισφορές ε, κτλ. Είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο προσλαμβάνουν τους ηλικιωμένους. Όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν ότι είναι πιστοί στους εργοδότες, ε, δεν ασθενούν, δεν απουσιάζουν, όλα αυτά δεν είναι σημαντικά. Το κόστος το εργασιακό είναι μικρότερο και γι' αυτό προσλαμβάνουν οι εργοδότες ηλικιωμένους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Αγουστίν, θα θέλατε να απαντήσετε. E, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια αντίφαση ανάμεσα σε αυτό και σε αυτό το οποίο είπα εγώ. Είπα ότι μετά από κάποιες πρώτες επιτυχείς προσπάθειες, ε, τώρα πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει και ο κόσμος μένει συνήθως μετά από κάποια ηλικία εκτός αγοράς εργασίας. Αναφέρθηκα επίσης και στα κίνητρα τα οποία θα πρέπει να δοθούν ιδιαίτερα στα πλαίσια της προσπάθειας για τη μείωση του κόστους της απασχόλησης. Ίσως τα κίνητρα αυτά να μην είναι επαρκή προς το παρόν. Ο στόχος του να παραμείνουν οι ηλικιωμένοι στην εργασία δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται δωρεάν. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Μπερές, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την Πολωνική Προεδρία για την πρόσκληση ε, που έκανε και σε εμά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα Κοινοβούλια των Κρατών Μελών να συζητήσουμε θέματα τα οποία δυστυχώς θα έλεγα ε, σήμερα παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για ε, τον κύριο Σεβερίν, επιμείνατε στο θέμα της εκπαίδευσης και νομίζω ότι αυτό έχει μεγάλη σημασία και τις σχέση της εκπαίδευσης με τη γύρανση του πληθυσμού και του σεβασμού που οφείλει η κοινωνία στους μεγαλύτερους στην ηλικία. Γίνονται πολλές συζητήσεις για τα συμβόλαια τιμής ανάμεσα στις γενναίες, για την αλληλεγγύη τη διαγενειακή και αυτό μάλιστα σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ήθελα να συνδέσω τη συζήτηση που κάνουμε σήμερα το πρωί με την καθημερινότητα των ευρωπαϊκών διαπραγματεύσεων και με τις συζητήσεις τις οποίες θα κάνουμε τους επόμενους μήνες οι οποίες μάλιστα εν μέρη έχουν ξεκινήσει γύρω από το θέμα των μελλοντικών δημοσιονομικών προοπτικών. Πολλές φορές στα πλαίσια της πολιτικής ζωής κάνουμε μεγάλες συζητήσεις ρητορικού και λυρικού πολλές φορές περιεχομένου. Αλλά όταν τα πράγματα επιστρέφουν στην πραγματικότητα, η εφαρμογή όλων αυτών των διακηρύξεων είναι κάτι το πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς λοιπόν σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εσείς σαν Κοινοβούλια των κρατών μελών το θέμα που μας απασχολεί σήμερα δεν μπορούμε παρά να το συζητήσουμε. Οι μελλοντικέ συζητήσεις για τις δημοσιονομικές προοπτικές είναι ένα happening ουσιαστικά στο Συμβούλιο που τελειώνει πάρα πολύ αργά με διακοπές επανειλημμένες, κραυγές, κλαφμούς πολλές φορές και νομίζω ότι και του χρόνου τα ίδια θα ζήσουμε. Θα πρέπει όμως εμείς σαν κοινοβούλια να είμαστε κάπως πιο ψύχρεμα γύρω από την υπόθεση αυτή. Υιοθετήσαμε κατά την αρχή της παρούσης κοινοβουλευτικής περίοδου τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Και όλοι συμφωνούμε για να πούμε ότι η στρατηγική αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική και σε σχέση με την λήψη υπόψη των δημογραφικών προκλήσεων που μας ενδιαφέρει σήμερα. Αν πιστεύουμε ότι η στρατηγική αυτή είναι καλή, το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να την χρηματοδοτήσουμε. Διαβλέπω εδώ ένα κίνδυνο. Πιστεύω ότι σε εθνικό επίπεδο οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων μας εξηγούν και μας λένε ότι τα πράγματα είναι πολύ οξυμένα. Είναι κατεπήγον να λύσουμε το θέμα του δημοσίου χρέους, Οπότε στο συγκεκριμένο αυτό πλαίσιο, στη συγκεκριμένη προσπάθεια δεν μπορούμε να βρούμε επιπλέον προϋπολογισμούς για τέτοιου είδους στόχους. Η αντίδραση δηλαδή σε αυτά τα οποία ζητάμε είναι εχθρική. Αν πράγματι όμως αυτό θέλουμε εμείς να κάνουμε, τότε οι στόχοι που έχουμε για τη συνοχή, για την αλληλεγγύη, τη διαγενειακή, οι προσπάθειες υπέρ της καλύτερης εκπαίδευσης που είναι ο καλύτερος τρόπος για την Ένωση να αντιμετωπίσει την πρόκληση της παγκοσμιοποίησης. Αν δεν κάνουμε σωστά ό,τι πρέπει τότε θα χάσουμε σε όλα. Πρέπει να είμαστε λοιπόν θαραλέοι και να πούμε ότι ακριβώς το πλαίσιο αυτό πρέπει να πατάμε καλά στο χώμα. Πρέπει από τη μία να προσπαθήσουμε φυσικά να αποκαταστήσουμε τους, ε, τα, τα, τα δημόσια λογιστικά, να ελαφρύνουμε την πίεση, εν πάση περιπτώσει, του δημοσίου χρέους, αλλά ταυτόχρονα να επενδύσουμε και στο μέλλον. Και αυτό θα γίνει και μέσω του προϋπολογισμού το, της Ένωσης και μέσω του προϋπολογισμού των κρατών μελών συνέργεια ανάμεσα στα δύο. Πρέπει λοιπόν να μας στηρίξετε έτσι ώστε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ισχυρό γιατί τότε μόνο θα μπορέσουμε να πετύχουμε στους στόχους μας. Οπότε το θέμα είναι λοιπόν αν συμφωνείτε με την πρόταση αυτή και με ποιο τρόπο μπορούμε από κοινού να προχωρήσουμε. Πράγματι ακούγεται απλή η ερώτηση, θα δούμε τώρα στη συνέχεια τι απαντήσεις θα δοθούν. Ο κύριος Σεβερίνα. Έχετε απόλυτο δίκιο όταν λέτε ότι σε σχέση με την παρέμβασή μου υπήρξαν τοποθετήσεις ε, συλλήρδιν και είναι σαφές ε, ότι πρέπει να τονιστεί ότι η υλοποίηση αυτών δεν είναι ε, αυθύνη, είναι δαπανηρά όλα αυτά και θα κοστίσουν και στη συζήτηση για τα δημοσιονομικά και τους προϋπολογισμούς πρέπει να διαρωτηθούμε πώς αυτή οι οι προκλήσει αντανακλώνται στην στρατηγική για παράδειγμα τη Ευρώπη για το 2020 και πώ θα υλοποιηθούν όλοι αυτοί οι στόχοι, πώ θα επιτευχθούν. Πρώτα απ' όλα έκανα μια έκκληση που απίφθηνα σήμερα το πρωί εδώ ώστε τουλάχιστον να μην μειωθούν, να μην μειωθούν τα κονδύλια των ταμείων που στρέφονται στην επίτευξη των κοινωνικών στόχων όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, στόχους κοινωνικούς από πλευράς οικονομικής δράσης. Δεύτερον, πρέπει να τονίσουμε και να μην υπεκφύγουμε τη συζήτηση για την διασπάθηση κοινωνικών κονδυλίων, ε, κοινοτικών κονδυλίων. Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει, υπάρχει ο φόβος της διασπάθησης. Και εδώ έχουμε σημαντικότατους στόχους και όταν ε, ζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξεταστούν καλά οι στόχοι όσον αφορά τους ουσιοδέστερους στόχους που θα έχουμε ενώπιον μας, πρέπει να αφαιρέσουμε ό,τι δεν είναι αποτελεσματικό και λειτουργικό. Εμείς στο προηγούμενο πάνελ, στο προηγούμενο γύρο, κάναμε λόγο ότι όλα αυτά τα κονδύλια, τα, μεγάλα, τα πολλά ευρωπαϊκά κονδύλια δημιουργούν δεκάδες χιλιάδες, μυριάδες θέσεις εργασίας. Είναι σαφές ότι αν διαιρεθούν όλα αυτά τα κονδύλια δια του αριθμού των χωρών, τότε δεν είναι τόσο τεράστια και η αποτελεσματικότητα στον κοινωνικό τομέα μπορεί να διευρυνθεί και να αυξηθεί και μπορούμε να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί. Αυτό είναι ένα στόχο που πρέπει να έχουμε ενώπιον μα. Δεύτερον, είναι σαφέ φυσικά ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια κατάσταση ότι όταν υπάρχει αναζήτηση εξοικονομήσεων μπορούμε να βρεθούμε στο περιθώριο των στόχων που θέλουμε να επιτύχουμε με τη στρατηγική του 2020. Ακόμα θα μπορούσε να συμβεί και το εξή. Πρώτα απ' όλα να αναζητηθούν ε, εξοικονομήσεις και να αναζητηθούν στην κοινωνική πολιτική. Κάτι τέτοιο εγώ θεωρώ ότι όχι μόνο στις ευρωπαϊκές χώρες ε, πρέπει να αντιμετωπιστεί η απειλή της χρεοκοπίας που επικρέμαται ως δαμόκλειο σπάθη. Επίσης πρέπει να δούμε τις πιέσεις ε, και να αντιμετωπίσουμε την ε, απειλή αυτή και κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την απειλή μόνο του. Χρειάζεται η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η παρέμβαση και ο στόχος της παρέμβασής μου και ο στόχος αυτών που προανέφερα κυρία είναι ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε όλα όσα είναι σε ένα κοινοτικό πλαίσιο να τύχουν κοινοτικών ευρωπαϊκών λύσεων και να μην υπάρχουν κατακαιρματισμένες προσπάθειες. Ευχαριστώ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αγουστίν. Ο επόμενος αγορητής που ζήτησε να παρέμβει είναι ο κύριος Κέβιν Χόπκινς από την Βουλή των Κοινοτήτων από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Χαίρομαι για την ευκαιρία να παρέμβω πάλι και ευχαριστώ τον κύριο Αγουστίν για αυτήν την πολύ χρήσιμη εισαγωγή του. Συζητούμε εδώ το θέμα της αλληλεγγύης μεταξύ γενεών οι νεότεροι να υποστηρίζουν τους πιο ηλικιωμένους κτλ. Και προφανώς Θέλουμε περισσότεροι ηλικιωμένοι να απασχολούνται και να έχουν μια θέση εργασίας και περισσότερες γυναίκες, σίγουρα. Πρέπει να τονίσουμε όμως ε, ότι η ε, έννοια της πλήρους απασχόλησης, ε, η κατανομή λοιπόν που μπορεί να μην θεωρείται δίκαια μεταξύ νέων και ηλικιωμένων ή μεταξύ εκείνων που έχουν παιδιά που έχουν μεγαλώσει ήδη ενώ άλλες οικογένειες έχουν παιδιά ακόμα, που, δεν, ε, που βρίσκονται στην παιδική ηλικία. Πρέπει να δούμε αυτές τις διαφορές. Αν όλοι ε, θέλουμε να εργαζόμαστε σε ένα καθεστώς πλήρους απασχόλησης και πληρώνουμε τους φόρους ε, και τότε θα, θα υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης όλων των αναγκών. Όμως εδώ οι συνταξιοδοτούμενοι πρέπει να τύχουν και ειδική υποστήριξη. Η πλήρης απασχόληση λοιπόν είναι η έννοια που είναι το πρόβλημα εδώ και κατανέμουμε από το ένα τμήμα της ε, ζωής ε, των ανθρώπων ε, προς την άλλη ηλικιακή ομάδα. Θα μπορούσαμε έτσι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Πληρώνουμε για κοινωνικούς στόχους μιας κοινωνίας που αποτελούμε και εμείς τμήμα της. Και για παράδειγμα, όσον αφορά τις κρατικές συντάξεις και τις εθνικές εισφορές για το συνταξιοδοτικό σύστημα, μετά έχουμε και τις ε, ε, καλυπτόμενες με αυτόν τον τρόπο συντάξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αν εργάζεται κανείς ε, και πληρώνεται με αυτόν τον τρόπο, δεν θα, υπήρχε κάποια, δεν θα υπήρχαν παράπονα, διότι εμείς θα είμαστε εκείνοι που θα απολάμβαναν των ωφελημάτων στο τέλος τέλος. Αλλά πρέπει να δούμε αν ε, σε σχέση με την αλληλεγγύη κάτι τέτοιο μπορεί να λειτουργήσει. Αν είχαμε βέβαια πλήρη απασχόληση ή πλήρη απασχολησιμότητα. Δεν έχουμε όμως πλήρη απασχόληση ή απασχολησιμότητα. Πρέπει να είναι κύριος στόχος στις κοινωνίες μας σε διεθνές επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο αυτός ο στόχος. Και αν πράγματι βρούμε, και αυτή είναι η περίπτωση, ότι σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο, φιλελευθερωποιημένο, απελευθερωμένο στις συναλλαγές κόσμο, δεν παράγεται πλήρης απασχόληση παράγονται υψηλά επίπεδα ανεργίας και υπάρχουν πάρα πολλές ανισότητες επίσης που δημιουργούνται και αυτό δημιουργεί παράπονα όσον αφορά την πληρωμή φόρων και τις εισφορές κάτι το οποίο δεν είναι και πολύ καλό φαινόμενο και αυτό το αναφέραμε χθε. όταν υπάρχει υψηλό επίπεδο φορολογίας και υπάρχουν υψηλά επίπεδα αντισταθμίσεων που δίνονται σε εκείνους που πληρώνουν υψηλούς φόρους ε, δεν υπάρχει πρόβλημα στις σκανδιναβικέ χώρες είναι μια ακραία περίπτωση που είναι είναι μια πολύ επιτυχής μορφή κοινωνιών. Είχα πάει στη Δανία πρόσφατα την προηγούμενη εβδομάδα και είναι σαφής η αντίθεση. Δανίας ε, ε, Ηνωμένου Βασιλείου όπου με χαμηλή φορολογία που είχε ακολουθηθεί ως πολιτική υπήρχε μια διαφοροποίηση σε σχέση με αυτά που γίνονται στη Σκανδιναβία. Είναι για παράδειγμα ε, 3% ε, η φορολογική επιβάρυνση 200 δις ε, για παράδειγμα για μας αν ίσχυε κάτι τέτοιο ε, τεράστιο ποσό όλα αυτά όμως σε σχέση με, ένα, με μια δυνατότητα πλήρους απασχόλησης τονίζω ότι θα συνεχίσω να εξετάζω αυτό το θέμα ήμουν επικεφαλής της ομάδας που είχε δημιουργηθεί για την Βουλή των Κοινοτήτων για τα θέματα πλήρους απασχόλησης όταν έρχεται η ώρα να εξετάσουμε την περίπτωση των ηλικιωμένων εργαζομένων και εγώ ίδιος δεν είμαι πλέον πλέον τόσο νέος και έχω συμφέρον να το εξετάσουμε αυτό. Ακούσαμε για περιπτώσεις ε, που ε, απασχολούν κάποιοι ηλικιωμένου. Είναι ιδιαίτερα, θα έλεγα, συνειδητοποιημένοι, είναι ιδιαίτερα επιμελείς και με ζήλο εργαζόμενοι, έχουν ε, καλές επιδόσεις, είναι πιστοί, είναι πολλές φορές πάρα πολύ προνομιούχο το να μπορεί κανείς, είναι προτέρημα να απασχολεί κανείς ηλικιωμένους και ίσως θα ήθελαν να εργάζονται και για μερική απασχόληση, γιατί έτσι θα μπορούσαν να συμπληρώνουν το εισόδημά τους. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί ηλικιωμένοι που θέλουν να εργαστούν και δεν υπάρχουν θέσεις απασχόλησης για αυτούς. Και αυτό συμβαίνει και στην ε, Μεγάλη Βρετανία. Υπάρχει η λατρεία των νέων, της νεότητας. Θεωρούν όλοι ότι είναι πιο ελκυστικοί, πιο θελκτικοί οι νέοι για τους εργοδότες. Και όσον αφορά το θέμα της αξιοπιστίας, ε, η ε, αποτελεσματικότητας δεν νομίζω να συμβαίνει αυτό ως κριτήριο. Οι ηλικιωμένοι πρέπει να έχουν ευκαιρίες να απασχοληθούν, όπως και οι νέοι πρέπει να έχουν ευκαιρίες να εργαστούν και να απασχοληθούν θα πρέπει να εξεταστεί και να οικοδομηθεί η έννοια, να προσεγγιστεί και να επιτευχθεί η έννοια της αλληλεγγύης. Μεγάλωσα στην γενιά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπήρχε τότε αλληλεγγύη. Χάθηκε σήμερα αυτή η αλληλεγγύη. Εγκαταλείφθηκε και ε, ακολουθήθηκε διαφορετική πορεία, ίσως η δημοκρατική, θα έλεγα κοινωνία σε αυτή που μεγαλώσαμε εμείς ε, όταν είμαστε παιδιά. Σας ευχαριστώ κύριε Χόπκινς για την παρέμβασή σας. Πρωτού δώσω τον λόγο στον κύριο Αουγκουστίν να απαντήσει. Θα ήθελα να σας πω ότι η κυρία Εύα Κόπατς θα αναλάβει τώρα την Προεδρία. Είμαστε δύο συμπρόεδροι εδώ. Έχετε λοιπόν τον λόγο κυρία Αουγκουστίν. Ε, Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις που έκανε ο κύριος Χόπκινς. Θα ήθελα να σας πω το εξής ε, για αυτά τα θέματα. Ίσως σήμερα μέσω αυτού του ονείρου, του σοσιαλδημοκρατικού ονείρου για την πλήρη απασχόληση θυμόμαστε με αρκετή απόσταση και νοσταλγώντας ακόμα και όλα σε αυτή την προοπτική ως δυνατότητα. Δεν το έχουμε όμως αυτό μπροστά μας ε, ως ε, γεγονός, την πλήρη απασχόληση. Πρέπει να πούμε ότι η, η ερώτηση σε σχέση με τα ιδανικά τα θέματα που τίθενται όταν μιλάμε για ιδανικά Πάρα πολλά πρέπει να γίνουν γιατί υπάρχουν πάρα πολλά άτομα χωρίς ε, εργασία, χωρίς απασχόληση. Πώς θα διαχειριστούμε τα κράτη μας ώστε να μπορέσουν να δημιουργηθούν αυτές τις θέσεις απασχόλησης και να, λυθούν, να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και σε σχέση με τις δημογραφικές ε, απειλές που ε, διαγράφονται. Δεν υπάρχει μία και μόνη ενιαία λύση, είναι σαφές. Αλλά επίσης είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη δέσμευση, περισσότερες προσπάθειες από πλευρά των κρατών μας που πρέπει να γίνουν είναι σαφές ότι υπάρχουν διαφορετικές πορείες και προσεγγίσεις για τις οποίες έγινε λόγος. Πρώτον, κατάρτιση, εκπαίδευση, παιδεία, καλύτερη προετοιμασία για να εισέρχονται στην αγορά εργασίας τα άτομα, νέοι, γυναίκες, ηλικιωμένοι, όλοι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι ως κράτος, ως χώρα να μειώσουμε το κόστος εργασίας και την επιβάρυνση που συνεπάγεται η πρόσληψη αυτών των ανθρώπων για την αγορά εργασίας ώστε να καταφέρουμε να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας και να επανανταχθούν σε αυτήν. Σε κάθε μια από τις χώρες μας θα πρέπει να γίνεται ό,τι μπορεί να γίνει και ό,τι είναι εφικτό με τα μέσα και τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως ε, για παράδειγμα αναφέρθηκε και από πλευράς ε, παρεμβάσεως για την Πολωνία. Θα πρέπει να δώσουμε επαρκή προσοχή να απασχολούμε ή να υποστηρίζουμε κάποιες αγορές ή τομείς έγινε πριν ε, λόγος για την μεταρρύθμιση της κοινωνικής ε, προστασίας μακροπρόθεσμα. Να τα πάρουμε ένα προς ένα. Τα κονδύλια που δίνονται στα ιδιωτικά ταμεία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια αγορά που θα δημιουργούσε πολλές θέσεις απασχόλησης σε όλη την Ευρώπη, πανευρωπαϊκά να λάβουμε υπόψη ότι αυτά τα ιδρύματα ή αυτές οι ιδιωτικές εταιρείες και επιχειρήσεις θα μπορούσαν να δίνουν μια απάντηση. Αυτοί οι μακροχρόνια άνεργοι θα μπορούσαν να επανέλθουν στην αγορά εργασίας, να είχαν κάποιες δυνατότητες. Θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ ε, και για τη εκπροσώπηση της ε, κυρίας από το, ε, ε, τη Βουλή της Πολωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε που μου δίνετε τον λόγο να παρέμβω. Παρακολουθώ αυτή τη συζήτηση με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα ήθελα όμως να επικεντρωθώ σε ένα άλλο θέμα και να θίξω κάτι άλλο. Κάναμε λόγο και είναι και του σειρμού, είναι της μόδας για την ισότητα των φύλων, ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Για παράδειγμα και σε σχέση με την Πολωνία αναφέρθηκε ότι τα παιδιά γεννιούνται. Υπάρχουν περισσότερα παιδιά ε, στις χώρες εκείνες όπου η ισότητα των φύλων έχει προχωρήσει και έχουν και απασχόληση, εργασία γυναίκες και αυτό είναι σαφές για όλους. Για την ισότητα των φύλων πρέπει να δώσουμε βάση σε αυτό το θέμα και να το εξετάσουμε σε βάθος να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο ώστε οι γυναίκε να έχουν θέσει εργασία, να έχουν απασχόληση. Ένα από τα στοιχεία θα ήταν η δυνατότητα να συμβιβαστεί η οικογενειακή ζωή με την επαγγελματική ζωή. Αυτό μπορεί να γίνει με διαφορετικού τρόπου, διευκολύνοντα για παράδειγμα την πρόσβαση στην αγορά εργασία στην Πολωνία. Εγκρίναμε ένα νομοθέτημα στην Πολωνία όπου γίνεται λόγο για νέε μορφέ περίθαλψη και φροντίδα των παιδιών, των πιο μικρών παιδιών και ελπίζουμε και θα έχει αυτό όπως βλέπουμε και ελπίζουμε αποτελέσματα στην προσχολική εκπαίδευση για παράδειγμα να διευκολύνουμε με νηπιαγωγία ή παιδικούς σταθμούς να μπορούν οι γυναίκες να συνδυάζουν τον χρόνο εργασίας τους και να μπορούν και οι άνδρες να προσαρμόζονται σε αυτό το καθεστώς. Θέλω να κάνω λόγο για κάτι το οποίο είναι πιο δύσκολο να αλλάξει. Βρίσκεται στην οτροπία, στη σκέψη των ανθρώπων. Όταν κάνουμε λόγο για την ισότητα των φίλων οι γυναίκες, πώς να το πω, αντιμετωπίζονται σαν εκείνες που βρίσκονται πίσω ή από κάτω και ε, χωλένουν και πρέπει να βοηθηθούν. Οι άντρε και οι γυναίκε όμω πρέπει ισότιμα, με ίσο τρόπο, με ισοδίκαιο τρόπο να αντιμετωπίζονται. Γίνεται όταν γίνεται λόγο για υποχρεώσει ανδρών και γυναικών. Και οι γυναίκε να αντιμετωπίζονται όταν γίνεται λόγο για την οικογένεια και την εκπαίδευση και ανατροφή των παιδιών να έχουν ίσο ρόλο και να συμμετέχουν εξίσου. Σε πολλέ χώρε και στην Πολωνία λέγεται ότι η γυναίκα είναι εκείνη η οποία μεγαλώνει το παιδί και το ανατρέφει και είναι υπεύθυνη για τη ζωή του παιδιού. Η γυναίκα είναι εκείνη που είναι στο σπίτι, που προετοιμάζει τα περιθάλπη, φροντίζει το παιδί, τα παιδιά κτλ. Οι αλλαγέ που χρειάζονται χρειάζονται χρόνο για τις νοοτροπίες, για την αλλαγή νοοτροπίας. Πρέπει να δραχθούμε τη ευκαιρία. Υπάρχουν μέσα και μέσα και εργαλεία στι ευρωπαϊκέ χώρε για διαφορετικέ κοινωνικέ δράσει προ αυτόν τον στόχο. Αν δεν το κάνουμε, όσο καλέ και να είναι οι πολιτικέ λύσει, δεν θα αλλάξει η κατάσταση των γυναικών στην αγορά εργασία κυρίω. Ευχαριστώ. Κύριε Αγουστίν, έχετε τώρα τον λόγο να απαντήσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μπορώ να κάνω λόγο για τον πιγκουίνο. Πιγκουίνος που μπορεί να είναι ένα σύμβολο για την ισότητα των ανδρών και των γυναικών. Διότι αυτό το πουλί που δεν πετάει ο πιγκουίνος που είναι τόσο ευφιές ον φροντίζει τα παιδιά του, τους νεοσούς, τους, τους του που εκολάπτονται από τα αυγά και σε ένα ισότιμο πλαίσιο μεταξύ ε, θήλεων και αρένων. Είναι ένα καλό σύμβολο. Αυτό εδώ το μικρό πιγκουινάκι στο πέτο που μπορεί να είναι ένα σύμβολο για την ισότητα γενεών. Από τα στοιχεία αυτής της διάσκεψης υπάρχει μια σειρά μελετών που βασίζονται σε ε, αυτά ε, τα ε, βιώματα. Δείχνεται ότι είναι ένας μύθος ότι οι παραδοσιακές οικογένειες, εκείνες οι γυναίκες στις παραδοσιακές οικογένειες που διαδραματίζουν ένα παραδοσιακό ρόλο και ασχολούνται με τα οικιακά και τα οικογενειακά τους θέματα, σε, εκείνα τα παιδιά, σε εκείνες τις οικογένειες λέει γεννιούνται περισσότερα παιδιά καθόλου. Αν δούμε το χάρτη της δημογραφικής ανάπτυξης και γεννητικότητας στην Ευρώπη μπορεί να δει κανείς ότι μεγαλώνουν περισσότερες οικογένειες και τα παιδιά σε εκείνες τις χώρες όπου δεν διατηρούνται οι παραδοσιακοί ρόλοι για τους άνδρες και τις γυναίκες. Το αντίθετο συμβαίνει. Σε εκείνες τις χώρες όπου υπάρχει ισότητα ευκαιριών και ισότητα φύλων και υποστηρίζεται η ισότητα των γυναικών στην αγορά εργασίας και η απασχόληση των γυναικών, σε εκείνες τις χώρες γεννιούνται περισσότερα παιδιά και η γεννητικότητα βαίνει καλώς. Και τώρα, πέρα από το ότι συμβαίνει αυτό, ε, για τους γάμους που συνάπτονται έχουμε και περισσότερα διαζύγια σήμερα και πρέπει να δούμε πώς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και άλλες παραμέτρους και άλλα στοιχεία όταν θα γίνεται ε, λόγος για αυτή την πολιτική υπέρ των οικογενειών. Σας ευχαριστώ κύριε. Και τώρα θα λάβει τον λόγο ο εκπρόσωπος ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κυρία Μάισνερ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Θα μιλήσω στα γερμανικά, στη μητρική μου γλώσσα. Το θέμα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και γι' αυτό ζήτησα και εγώ τον λόγο. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω κάτι, κυρία Αουγουστίν, όσον αφορά την άποψη για την δημογραφική ανανέωση. Τέλεια ακούγεται αυτό. Και όλοι θα ευχόμαστε περισσότερα παιδιά να γεννιόντουσαν. Διότι ε, διαφορετικά θα έπρεπε να αναχαιτιστεί η δημογραφική εξέλιξη και βλέποντας ότι υπάρχουν περισσότερα παιδιά και πιο περισσότερες έγκυες γυναίκες. Ένα συγκεκριμένο στοιχείο γι' αυτό. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέρυσι μιλήσαμε για την γονεϊκή άδεια, την άδεια για τις μητέρες. Όταν γεννιέται κάποιο παιδί δεν είναι καθόλου κάποια ασθένεια, είναι όμως μια σημαντική τομή, μια καμπή στη ζωή μιας γυναίκας και έχει πάρα πολλά να κάνει πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο λοιπόν για την απόφαση ότι 20 εβδομάδες μητρική άδεια, γονεϊκή άδεια πανευρωπαϊκά στην Ευρώπη θα πρέπει να εγκριθεί με 75% κάλυψη ε, όσον αφορά τα έσοδα της γυναίκας όμως ε, οι, τα οι χώρες πρέπει να μπορέσουν να προχωρήσουν είναι ωραίο να ζητάει κανείς μητρική άδεια, γονεϊκή άδεια με σχεδόν πλήρη, ε, πλήρης αποδοχές και να διασφαλίζεται η επιστροφή στο χώρο εργασίας και απασχόλησης των γυναικών. Ταυτόχρονα όμως οι εθνικοί, δημοσιονομ... τα... προϋπολογισμοί από τα κράτη-μέλη σε μια περίοδο κρίσης ε, συνεπάγονται περικοπές και πολιτική λιτότητας. Πώς μπορεί αυτό το... αυτή η αντίφαση να επιληθεί, αυτή η σύγκρουση αυτών των δύο στοιχείων να αντιμετωπιστεί. Έχετε κάποιο σχόλιο. Και το παράδειγμα με τον πιγκουίνο το βρήκα τέλειο. Πολύ ωραίο. Πραγματικά εν, μια κοινωνική αλλαγή χρειάζεται, μια κοινωνική μεταβολή. Εγώ είμαι μητέρα δύο παιδιών. Επτά μήνε απουσίασα από την απασχόλησή μου. Ο άντρα μου με υποστήριξε πλήρω και ο ίδιο επί ένα χρονικό διάστημα φρόντιζε τα παιδιά εκείνο. Για μένα δεν ήταν πρόβλημα το ότι εργαζόμουν για μισή μέρα μόνο, αλλά για τον άντρα μου ήταν πρόβλημα αυτό. Τώρα μεγάλωσαν τα παιδιά μα και έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Χρειάζεται μεγάλη μεταβολή, μεγάλη αλλαγή στι νοοτροπίε, στα μυαλά των των ανθρώπων προτού καταφέρουμε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους να έχουμε περισσότερα παιδιά. Το δεύτερο σημείο αφορά τους ηλικιωμένους εργαζομένους, τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Μιλήσατε για το πρόγραμμα για εκείνους που είναι 50 και παραπάνω, πιο μεγάλοι από τα 50 χρόνια στην Πολωνία. Θα ήθελα να ξέρω κάτι παραπάνω για αυτό το θέμα, για αυτή την πρωτοβουλία και δύο σχόλια από πλευράς μου. Το πρώτο, επισημάνατε ότι οι εργοδότες δεν προσλαμβάνουν με ιδιαίτερη ευχαρίστηση ηλικιωμένους. Ξέρουμε όμως ότι οι ηλικιωμένοι είναι πολύ πιο εύκολο και ε, λιγότερο δαπανηρό να φροντιστούν από ότι οι νεότεροι. Έχουν ήδη σταδιοδρομία πίσω τους, έχουν μεγαλύτερη πείρα, μπορούν πιο νυφάλια και με μεγαλύτερη σοφία και σύνεση να αποφασίζουν. Και είναι αυτό πολύ θελκτικό. Στη Γερμανία όμως υπάρχει μια σειρά εταιριών που υποδειγματικά είπαν ως πρότυπο ότι συνειδητά θα προσλαμβάνουμε ηλικιωμένους. Υπάρχουν και κάποιες εταιρείε που λένε ότι έχουν ένα πρόγραμμα πολυμορφίας, diversity program. Συνειδητά προσλαμβάνουν ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες ή με μειονεξίες. Και η πείρα δείχνει ότι είχαν δίκιο και δείχνει ότι η εμπειρία αυτή στέφθηκε με επιτυχία. Υπήρξαν επιτυχίες λοιπόν. Χρειαζόμαστε best practices, βέλτιστες πρακτικές που θα μας οδηγήσουν μπροστά. Και κάποιοι θέλουν περισσότερο να εργαστούν στη Γερμανία και όχι μόνο μέχρι το όριο ηλικίας συνταξιοδότησής τους. Και κάποιος ο οποίος μπορεί να εργαστεί και σωματικά περισσότερο θα μπορούσε αυτό να οδηγήσει στην εξοικονόμηση κονδυλίων. Δεν θα έπρεπε να παίρνουν χρήματα ως άνεργοι αυτοί οι άνθρωποι αν δεν είχαν μια θέση απασχόλησης. Μπορεί λοιπόν να είναι και φθηνότερη αυτή η λύση προσλαμβάνοντας ηλικιωμένου. Καλό θα ήταν αυτό να το λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο εκπρόσωπος του Βελγίου, ο κύριος Χέρμαν Τρόπερα, παρακαλώ. Ε, ομολογώ ότι είμαι διστακτικός ε, μπροστά σε αυτή την έκκληση περί ενθάρρυνσης κάποιων δημογραφικών τάσεων. Παράδειγμα, η Κίνα. Η Κίνα ένα δις 300 εκατομμύρια κατοίκων με μια πολιτική αντίθετη με τις δημογραφικές εξελίξεις. Ένα παιδί ανά νοικοκυριό στην Κίνα δημιουργεί τώρα ή σε λίγα χρόνια εκατοντάδες εκατομμύρια ηλικιωμένων. Λοιπόν, πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στην Κίνα με 300 εκατομμύρια συνταξιούχων που δεν αντικαθίσταται από ένα παιδί. Γιατί φυσικά ένα στα τέσσερα δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες. Δεύτερη παρατήρηση. Στις δικές μας χώρες, στα πιο φτωχά νοικοκυριά, έχουμε τα περισσότερα παιδιά. Στις Βρυξέλλες, σαν παράδειγμα, το πρώτο όνομα των παιδιών δεν είναι Πιέρ, δεν είναι Ζω, αλλά Μοχάμεντ. Αυτό σημαίνει ότι οι οικογένειες, τις οποίες σέβομαι ιδιαιτέρως και που έχουν μια μικρή προσαρμοστικότητα στις κοινωνικές πιέσεις, διατηρούν μια δημογραφική συμπεριφορά με περισσότερα παιδιά από ότι ο μέσος όρος. Ε, παράδειγμα, η Ρώμα από τη Βουλγαρία, από τη Ρουμανία, από άλλες χώρες της κοινότητας δημογραφικά συμπεριφέρονται ε, με πάρα πολλά παιδιά ενώ δεν προέρχονται από υψηλά οικονομικά στρώματα. Πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε σε ποια πλευρά βρίσκονται οι λεγόμενες δημογραφικές δεξαμενές. Τελευταία παρατήρηση για τους λιγότερο ε, νέους εργαζομένους. Αποφασίστηκε στο Βέλγιο ότι οι συνταξιούχοι μπορούν χωρίς όριο να δουλεύουν αν θέλουν, να κερδίζουν αν θέλουν. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι περιορισμοί ε, φορολογικοί, αλλά δεν υπάρχει απαγόρευση του να δουλεύει κανείς μετά από την ηλικία συνταξιοδότητης χωρίς να χάνει φυσικά τη σύνταξή του. Και αυτό είναι μια δυνατότητα την οποία θα πρέπει να εξετάσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει μία μπλε κάρτα. Η πρόεδρος, αν θα ήθελε να κάνει κάποια παρατήρηση σε σχέση με την τελευταία παρατήρηση που έγινε από τον Βέλγο εκπρόσωπο. Ναι, ευχαρίστω. Μπορώ να το κάνω. Δεν θεωρώ ότι εγώ είμαι υπεύθυνη να απαντήσω, αλλά φυσικά πρόσεξα την ερώτηση και αναφέρθηκαν προγράμματα πολυμορφοποίησης, diversity programs ως παράδειγμα. Θεωρώ ότι αφενός χρειάζονται κίνητρα για τους ηλικιωμένους. Για παράδειγμα, σε σχέση με το Βέλγιο να υπάρχουν κίνητρα οικονομικά κίνητρα. Αυτό είχα αναφέρει, να υπάρχουν κίνητρα για εργαζόμενους και εργοδότες. Το άλλο που αναφέρατε, πρέπει να σκεφτούμε πού γεννιούνται τα παιδιά ακριβώ. Δεν συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά που γεννιούνται στην Ευρώπη είναι ευπρόσδεκτα. Αν μια οικογένεια δεν είναι ολοκληρωμένη στην κοινωνική ένταξη, πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να ενταχθεί κοινωνικά σε αυτή την ολοκλήρωση. Και τα, παιδιά, τα ζευγάρια ε, οι άντρες και οι γυναίκες ε, ε, πρέπει να μπορούν τα ιδανικά τους να τα υλοποιήσουν ώστε να αποκτήσουν οικογένεια. Οι γυναίκες όταν εργάζονται για παράδειγμα να μπορούν να συμβιβάσουν τις, τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις με την οικογένεια. Αυτό πρέπει να είναι ένας στόχος. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αγκουστίν, κύριε Γερουσιαστά, θέλετε να πείτε κάτι εσείς. Ευχαριστώ. Μάλιστα, κατά πρώτο λόγο στις παρατηρήσεις που έκανε η κυρία Πρόεδρος Μάισνερ θα ήθελα να αναφερθώ και να πω κάτι. Είναι σαφές ότι οι απουσίες όσον αφορά την ε, γέννηση ενός παιδιού ε, σε σχέση με την μητέρα όσον αφορά την εργασία της ε, όταν κάνω λόγο εννοώ για την άδεια τη γονεϊκή που εγκρίθηκε για τις γυναίκες όταν γεννούν παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και για την Πολωνία πρέπει να υλοποιηθεί αυτή η οδηγία αλλά για τη συζήτηση που έγινε είδαμε πώς υπάρχουν δικαιώματα για την άδεια γυναικών ε, να εγκαταλείψουν τη θέση τους απασχόλησης και να ασχοληθούν με τα παιδιά τους. Πρέπει αν ισχύουν μόνο για τις γυναίκες αυτά, δεν θα εξυπηρετηθούν οι γυναίκες όπως θα έπρεπε. Θα προσλαμβάνουν όπως επιθυμούν τους εργαζόμενους οι εργοδότες. Και γι' αυτό πρέπει να το δούμε αυτό και στην Πολωνία και σε άλλες χώρες. Αυτή η ευκαιρία να χρησιμοποιείται η απουσία της γυναίκας από το χώρο εργασίας λόγω γέννησης ενός παιδιού ή η γονεϊκή άδεια πρέπει να είναι η ίδια στο χαρακτήρα της και για τις γυναίκες και για τους άνδρες, για τους πατέρες και τις μητέρες και για μετά από τη γέννηση να μπορεί να ασχολείται η γυναίκα με την ανατροφή των παιδιών και πολλοί Πολωνοί θα ήθελαν να χρησιμοποιείται αυτή η γονεϊκή άδεια, η πατρική άδεια δεν θα έπρεπε τότε ο εργοδότης να επιλέγει μόνο άνδρες και όχι γυναίκες επειδή θα μπορούσαν οι άνδρες να παραμένουν διαρκώς στο χώρο απασχόλησης όταν γεννιέται ένα παιδί. Όταν ισχύει το ίδιο εξίσου για γυναίκες και άνδρες τότε και οι γυναίκες και οι άνδρες θα ωφεληθούν εξίσου. Και για το πρόγραμμα αυτό στην Πολωνία τρία στοιχεία έχει. Πρώτα απ' όλα να μειωθούν τα εργατικά κόστη, η εργασιακή επιβάρυνση. Πρέπει να πληρώνται λιγότερο περισσότερες εισφορές ε, όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, τα ταμεία εργασίας, ε, αν προσλαμβάνονται άτομα τα οποία έχουν πάνω από 50 ε, χρόνια ηλικιακά. Δεύτερο θέμα, η εκπαίδευση, παιδεία, κατάρτιση. Οι ηλικιωμένοι λοιπόν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα ευρύ φάσμα, ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών που στοχεύουν στην ενεργοποίηση ακριβώς στην αγορά εργασίας για αυτούς αν οι νέοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητες όσον αφορά την κατάτηση και εκπαίδευση, τότε θα ήταν σε, ε, θέση μειονεκτική ηλικιωμένη. Πρέπει όμως να δούμε ότι και οι ηλικιωμένοι ακριβώς μπορούν να υποφεληθούν με μαθήματα, ε, δυνατότητα επιμόρφωσης, κατάρτισης. Τρίτο, η πρόσληψη των ηλικιωμένων μέσω γραφείων ε, ξέβρεσης εργασίας μέσα στο πλαίσιο των κοινωνικών μέτρων υποστήριξης υπάρχει δυνατότητα να υπογραφούν συμβάσεις ώστε να ενεργοποιηθεί περισσότερο η πρόσληψη των ηλικιωμένων, να ενεργοποιηθεί αυτό το, αυτό το σκέλος στην αγορά εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται αυτό μέσω τέτοιων γραφείων και όχι μόνο μέσω των εθνικών γραφείων ε, εργασίας. Έχουμε ένα ποσοστό που είναι σημαντικό για την πρόσληψη των ηλικιωμένων με αυτόν τον τρόπο. Τώρα φυσικά με την κρίση δημιουργούνται νέα εμπόδια και νέα προβλήματα

Πρέπει να δούμε ότι είναι ευάλωτα αυτά τα ε, μέσα μέτρα και θα πρέπει να δούμε την πτυχή απώλειας θέσης απασχόλησης από τους ηλικιωμένους δεδομένης της κρίσης. Πρέπει όμως να αντιμετωπιστεί και αυτή η παράμετρος. Τώρα θέλω να στραφώ σε αυτό το οποίο είπατε για το ότι οι ηλικιωμένοι συνήθως θέλουν να εργαστούν περισσότερο από το όριο συνταξιοδότησής τους. Αληθεύει αυτό. 80% στην Πολωνία των Πολωνών θέλουν, ε, ονειρεύονται ότι θα μπορέσουν να ε, συνταξιοδοτηθούν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουν να εγκαταλείψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Και εκείνο για το οποίο πρέπει να, σε αυτό που πρέπει να επικεντρωθούμε είναι το εξής αν θέλουμε να περάσουμε από τη συνταξιοδότηση και ανάληψη νέας θέσης απασχόλησης ώστε να έχουμε δύο εισοδήματα από τη σύνταξη και από τη νέα δυνατότητα απασχόλησης. Δεν πρέπει να ε, τα απορρίψουμε αυτά ή να τα υποβαθμίσουμε. Πολλά άτομα που εργάζονται όσον αφορά τις υπηρεσίες ή την φροντίδα, την περίθαλψη, φροντίζουν παιδιά ηλικιωμένους. Υπάρχει όμως και μια φαιά ζώνη, μια γκρίζα ζώνη της παραοικονομίας. Η κυρία Πομάσκα και εγώ προσπαθούμε αυτά τα άτομα να περάσουν από τη φαιά γκρίζα ζώνη της παραοικονομίας στην επίσημη θεσμοθετημένη νόμιμη οικονομία και να μην εργάζονται στο πλαίσιο της παραοικονομίας και ξεκινά να λειτουργεί καλά αυτό αλλά για να μπορέσουμε να το πετύχουμε πρέπει να υπάρχει δέσμευση της, ε, του κράτους, του δημοσίου <clears throat> για την ε, κάλυψη εισφορών και ίσπραξη των ε, ε, πληρωμών και εισφορών. Πολλές φορές θέλουν να εργαστούν τα άτομα αυτά περισσότερο. Δεν είναι μόνο τα χρήματα, αλλά η δυνατότητα να συμμερίζονται αξίες και αρχές με άλλους ανθρώπους σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους ηλικιωμένους, είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για αυτούς. Θα ήθελα να σας πω επιπλέον και κάτι άλλο και αναφέρομαι εδώ σε αυτό το οποίο ανέφερε ο Βέλγος συνάδελφος, ο κύριος Δεκλό, στο ότι δηλαδή θα πρέπει, θα έπρεπε η Κίνα, την Κίνα να εξετάσουμε όταν κάνουμε λόγο για το ζήτημα της πολιτικής της δημογραφικής ανανέωσης όπου υπάρχουν ε, προβλήματα ή επιφυλάξεις. Προσέξτε, για τη Βουλγαρία ή η Ρουμανία για την γεννητικότητα, για το ανώτερο επίπεδο εκείνο το οποίο σημειώνουν από πλευράς γενετικότητας. Όμως ε, δεν μπορεί να θεωρηθεί μόνο πανάκια αυτό για την ανανέωση των γενεών βλέπουμε ότι έχουμε την κατάσταση στην Ευρώπη της δημογραφικής συρρήκνωσης. Θα έχουμε σε λίγα χρόνια ακόμα λιγότερους Ευρωπαίους. Θα υπάρξει αρνητική φθήνουσα εξέλιξη και πρέπει να δοθεί υποστήριξη λοιπόν στην, γενετική, στην γενεαλογική ανανέωση και αντικατάσταση των ε, γενεών και θα πρέπει να δούμε και το θέμα των μεταναστών που έρχονται σε εμά. Υπάρχουν Δαπάνε που εξαρτώνται από όλα αυτά. Θα πρέπει να επενδύσουμε ώστε οι Ευρωπαϊκέ οικογένειε να γεννούν παιδιά και αυτό θα δημιουργούσε λιγότερα προβλήματα και θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είδα μια μπλε κάρτα. Ο κύριος Ταντέουσον Τομασεύσκη έχει το λόγο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόεδρε, μία ερώτηση προς τον γερουσιαστή Ογκοστίν. Ε, σήμερα, όταν μιλάμε για την προπτική της ε, πιο μακρόχρονης παραμονής ε, στην αγορά εργασίας των ηλικιωμένων, πρέπει να δούμε και την πραγματικότητα, την δύσκολη οικονομική κατάσταση, τις περικοπές στον προπολογισμό, τις δημοσιονομικές δυσκολίες. Να δούμε ποιοι είναι οι άνεργοι ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νέοι αλλά και ηλικιωμένοι πάνω από τα 50. Εδώ ε, πρόκειται για ένα δίλημα. Και συμφωνώ εδώ με τον ε, γερουσιαστή. Δεν θα πρέπει να μειώσουμε τα κονδύλια προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά να αυξήσουμε τις προπτικές επενδύσεων για να αυξήσουμε τις θέσεις απασχόλησης και να τις μοιράσουμε μεταξύ των νέων και των ε, πάνω από 50. Ένα άλλο πρόβλημα αφορά στη συμμετοχή των, του κράτους ε, και των ευρωπαϊκών κονδυλίων ε, στην κατεύθυνση μιας καλύτερης προσαρμογής των ηλικιωμένων για να αντιμετωπίσουν ε, τις ε, προκλήσεις του σύγχρονου πολιτισμού και της σύγχρονης οικονομίας. Στην Ήπεθρο το πρόβλημα είναι ακόμη πιο αισθητό και εκεί πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα, ούτω ώστε όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να επανέλθουν στην αγορά εργασίας και πολλοί δεν το κάνουν γιατί ακριβώς δεν έχουν προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα στις νέες τεχνολογίες. Χρειάζεται λοιπόν βοήθεια, όχι μόνο εκ μέρους των κρατών μελών αλλά και των ε, Ευρωπαϊκών Ταμείων. Ευχαριστώ κύριε Τομασεύσκη, ο κύριος Αουγκοστίν. Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα την ε, λογική της ερώτησης του κυρίου Τομασεύσκη. Και στην Πολωνία περνάμε μια δύσκολη στιγμή κρίσης. Σε πολλούς τομείς θα πρέπει να περικόψουμε τη χρηματοδότηση για να επανεξισορροπήσουμε τον προπολογισμό μας. Γι' αυτό θα πρέπει να συγκεντρωθούμε στα πράγματα εκείνα τα οποία είναι πραγματικά θεμελιώδη. Απ' την άλλη, δεν στέκει ε, να, χρημα... να χρηματοδοτούμε τεράστια ποσά για την κάλυψη των ανέργων αλλά δίνοντάς τα στους εργοδότες. Από μόνο του το μέτρο της επανένταξης δεν αρκεί. Στην Πολωνία, στην Πολωνία Πολλές φορές έχουμε επενδύσει κεφάλαια στην αγορά εργασίας και όταν ε, χρηματοδοτήσαμε αυτά τα ποσά, μας είπαν οι εργοδότες θέλουμε και διευκολύνσεις, χωρίς διευκολύνσεις δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά τελικά τα άτομα με προβλήματα θα πρέπει να είναι αυτά τα οποία θα λαμβάνουν τη βοήθεια στις ε, περικοπές τώρα. Η Ευρώπη φωνάζει πειθαρχία, πειθαρχία, πειθαρχία και ε, πρόκειται για τον όρο που είναι της μόδας σήμερα. Φυσικά, συμφωνώ, θα πρέπει να πειθαρχήσουμε και να πειθαρχήσουμε και τις κοινωνικές δαπάνες. Εκείνες οι οποίες συνδέονται με δημογραφικά ζητήματα χρειάζεται μεγαλύτερη πειθαρχία και στην πολιτική αλληλεγγύης. Απ' την άλλη μεριά όμως υπάρχουν και όρια και αυτοί που φτιάχνουν τον προϋπολογισμό θα πρέπει να θυμούνται ότι η πολιτική της πειθαρχία δεν θα πρέπει να ξεχάσει εντελώς τι είναι πειθαρχία. Η αλληλεγγύη είναι μία από τις πιο σημαντικές ιδέες που πρεσβεύουμε όχι μόνο στην Πολωνία αλλά και στην Ευρώπη αλληλεγγύη μεταξύ νέων και ηλικιωμένων, ηλικιωμένων προς τους νέους. Θα έπρεπε λοιπόν αυτή η αλληλεγγύη μεταξύ των γενιών θα πρέπει να βοηθιέται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίοδο κρίσης. Πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τους πιο σημαντικούς στόχους. Ευχαριστώ κύριε Γερουσιαστά. Μια μπλε κάρτα. Σας δίνω το λόγο, αλλά παρακαλώ συστηθείτε. Σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να πω ότι συμφωνούμε ότι οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να βρουν τη σωστή θέση τους στην αγορά εργασίας. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι δεν υπάρχουν αυτές οι θέσεις στην αγορά εργασίας. Και δεν είναι η πραγματικότητα ότι αν επιλέξουμε ένα άτομο, αν δημιουργήσουμε μια προτιμησιακή, ένα προτιμησιακό καθεστώς ε, για κάποια άτομα στην αγορά εργασίας, τότε αυτό γίνεται εις βάρος κάποιων άλλων. Λυπάμαι, ίσως είμαι είναι πολύ ρεαλιστική, πραγματιστική αυτή η προσέγγιση, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην Εστονία, για παράδειγμα, έχουμε πολλούς νέους. Νέους ανθρώπους που είναι μακροχρόνια άνεργοι. Και πολύ προσωπικά μια παρατήρηση. Ο μεγαλύτερος γιος μου είναι 22 ετών. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο ε, δευτεροβάθμιο επίπεδο και πάρα πολλοί βρίσκονται άνεργοι από τους συμμαθητές του, έχουν εγκαταλείψει υπάρχει εγκατάλειψη και δεν υπάρχει προοπτική να απασχοληθούν. Και αυτό συμβαίνει για πολλούς ε, μακροχρόνια άνεργους. Και αυτό τώρα για τους πιγκουίνους. Εγώ είμαι γυναίκα, έχω παιδιά. Θα έλεγα ναι, θα έπρεπε όλοι να έχουν ίσες ευκαιρίες σίγουρα ε, μπαίνοντα ή έχοντας προσπελασιμότητα πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Όμως δεν υπάρχουν και τόσες πολλές θέσεις εργασίας, τουλάχιστον στην Εστονία. Υπάρχουν κάποιοι τομείς, συγκεκριμένοι κλάδοι, όπου το χάσμα είναι 33% μεταξύ γυναικών και ανδρών. Οι γυναίκες υποχρεούνται να το δεχθούν αυτό το μισθολογικό χάσμα, αυτό τη μισθολογική διαφορά. Το λέω αυτό επειδή το ξέρω. Όταν υπάρχουν συνεντεύξεις ε, για την πρόσληψη υπάρχει η ετοιμότητα ε, η προθυμία να προσαρμοστούν με αυτόν τον τρόπο αναγκαστικά σε αυτές τις διαφορές. Και μια άλλη τάση, θλιβερή και αυτή, αξιολύπητη, η ρωσική μειονότητα, οι ηλικιωμένοι άντρες από αυτούς είναι άνεργοι, χωρίς να μπορούν να απασχοληθούν. Πολλές φορές οι γυναίκες τους έχουν δύο ή τρεις εργασίες, εργάζονται δύο, σε δύο ή τρεις εργασίες οι άντρες ε, απλά ξαπλώνουν στα, στους καναπέδες και παρακολουθούν ποδοσφαιρικούς αγώνες και βρίσκονται και όλο σε μεγαλύτερη απόγνωση και απογοήτευση. Είναι πολύ περίπλοκο το θέμα. Ερώτηση. Ποια είναι η προτεραιότητα που έχετε για την αγορά εργασίας. Θα έπρεπε να είναι ηλικιωμένοι ή όχι και με ποιες επιπτώσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Τώρα ο κύριος Αυγουστίν nie Κύριοι, μην ξεκινήσουμε πόλεμο μεταξύ των γενιών ε, για την κατάκτηση μιας θέσης εργασίας. Οι μελέτες στην Ευρώπη αποδεικνύουν ότι Οι περισσότεροι άνεργοι βρίσκονται στις περιοχές εκείνες όπου έχουμε και τη μεγαλύτερη ανεργία ηλικιωμένων. Η ανεργία των ηλικιωμένων δεν ευνοεί την απασχόληση των νέων. Το αντίθετο. Οι κατάλληλες πολιτικές για τους ηλικιωμένους διευκολύνουν και στη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους και μειώνεται και η πίεση στο κόστος εργασίας. Στοιχίζει πάρα πολύ το να διατηρούμε τους ηλικιωμένους σε κατάσταση παινίας. Διότι κάποιος πρέπει να καταβάλει αυτά τα χρήματα για την παροχή υπηρεσιών. Τώρα αν εργάζονται, αυξάνονται και τα κονδύλια εκείνα υπέρ των ταμείων και υπέρ της ανάπτυξης. Παράδειγμα, Πολωνία. Εδώ έχουμε και υπουργού που μπορούν να με διορθώσουν αν θέλουν. 94 εκατομμύρια σλότη θα πρέπει να καταβάλουμε φέτος για να καλύψουμε τα κενά των ταμείων. Αν αυτά τα σλότη τα επενδύαμε αλλού, θα είχαμε πάρα πολλές θέσεις, νέες, νέες θέσεις εργασίας στην Πολωνία. Αυτό όμως δεν το κάνουμε. Και το επίπεδο ανεργίας είναι πανύψηλο. Και μεταξύ των νέων και μεταξύ των ηλικιωμένων. Γι' αυτό η αηφορία του προϋπολογισμού και των συνταξιοδοτικών ταμείων είναι σημαντική και για τους νέους και για τους ηλικιωμένους. Εργαζόμενοι ηλικιωμένοι δεν αφαιρούν δουλειά από τους νέους. Όταν εργάζονται παραπάνω οι ηλικιωμένοι βοηθούν τους νέους και θέλω να το τονίσω αυτό. Πράγματι οι διαφορές αμοιβών μεταξύ νέων και γέρων είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Είναι άνισες. Δεν θα έπρεπε να έχουν έτσι τα πράγματα και αυτό για διάφορους λόγους. Όχι μόνο για το λόγο του θέματος των διακρίσεων, αλλά αλλά συχνά οι γυναίκες έχουν λιγότερη κινητικότητα, άρα αμείβονται λιγότερο. Ναι, υπάρχει πρόβλημα διάκρισης μεταξύ των μισθών ανδρών γυναικών. Ένα φαινόμενο το οποίο θα πρέπει να το καταπολεμήσουμε αποφασιστικά. Στο Πολωνικό Κοινοβούλιο έχουμε μία ομάδα γυναικών η οποία ολοένα και μεγαλώνει η οποία ετοιμάζει ένα πακέτο πρωτοβουλειών για να πείσει τους εργοδότες να αντιμετωπίζουν ισότιμα τους άντρες και τις γυναίκες στον τόπο εργασίας. Κυρίως όταν ε, ε, έχουμε προσλήψεις σε θέσεις υψηλού επίπεδου και φυσικά θα, δώσουμε και θα βοηθήσουμε και εμείς αυτήν την ομάδα. Η κυρία Μπιλιέτα από το Μαλτικό Μαλτέζικο Κοινοβούλιο θέλει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολλές συζητήσεις γίνονται για την απασχολησιμότητα ηλικιωμένων ατόμων. Και όπως είπε ο γερουσιαστής Αυγουστίν, δεν είναι δίλημα μεταξύ γενεών. Όμως συμφωνώ με, το, με την εκπρόσωπο από την Εστονία. Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τους νέους έχει ακόμα πιο κέρια σημασία. Δεν σε σχέση με τις ε, βλέψεις που έχουν ή την επιθυμία τους να δημιουργήσουν ε, οικογένεια, αυτές δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν αν είναι άνεργοι. Θα πρέπει να δούμε, ακόμα και αν διατηρήσουμε τις ε, βιομηχανικές μας δράσεις, θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικές ε, με τη χρήση αυτοματισμού, με τη χρήση δηλαδή ε, ρομπότ και μηχανών και έτσι όλο και λιγότεροι εργαζόμενοι, λιγότεροι άνθρωποι θα χρειάζονται. Έχουμε προβλήματα λοιπόν σε σχέση με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης για την μετάθεση ε, όσον αφορά τα επιδόματα ανεργίας και τη μείωση της επιβάρυνσης δημιουργώντας και νέες θέσεις απασχόλησης όσον αφορά και τον κοινωνικό τομέα. Αυτό θα ήθελα να θέσω σε ερώτημα στον Γερουσιαστή Αγγουστίν. Τι θα λέγατε γι' αυτό, Γερουσιαστή Αγγουστίν να μεταθέσουμε αυτή την ε, νοοτροπία του όλο και περισσότεροι νέοι να είναι στην ανεργία και να μπορέσουν με κάποιο τρόπο να είναι απασχολήσιμοι και να εργαστούν, παρότι μπορεί να μην είναι απόλυτα παραγωγική η εργασία τους. Θα δοθεί όμως η πείρα, η εμπειρία σε αυτούς τους νέους ανθρώπους που θα ενδυναμώσει την αγορά εργασίας μακροπρόθεσμα και θα οδηγήσει σε νέες ευκαιρίες δημιουργίας θέσεων απασχόλησης μακροπρόθεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ και στη συνέχεια η κυρία Μαζούρεκ θα λάβει τον λόγο βουλευτής στην ε, Πολωνική Εθνοσυνέλευση. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ προσθέτω τη φωνή μου σε αυτά και θέλω να αναφερθώ στην απάντηση που έδωσε πιο πριν ο κύριος Αγουστίν σε σχέση με το ότι οι γυναίκες δεν, δεν έχουμε τέτοια κινητικότητα. Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό. Είμαστε εξίσου εύκολα, ε, μπορούμε εύκολα να κινηθούμε και να μετακινηθούμε και να προσαρμοστούμε όπως ε, οι άνδρες. Και σε σχέση και με τις μισθολογικές διαφορές που υπάρχουν διεκδικούμε την ισότητα των μισθών. Και σε σχέση για την διαφοροποίηση όσον αφορά την απασχόληση για τους νέους και ηλικιωμένους Πρέπει να βρεθούν τα μέσα και εργαλεία ώστε να μπορέσουν οι εργοδότες να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας ειδικά για τους νέους αλλά και για τους ηλικιωμένους. Για μας όμως το πιο σημαντικό για το Εθνικό Κοινοβούλιο αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε να τηρούμε και να συμμορφωνόμαστε με την ομοθεσία κανονισμούς και οδηγίες για να είναι αποτελεσματικοί αυτοί οι νόμοι και να βρεθούν απαντήσεις στις ανάγκες το αν δεν είναι αποτελεσματικοί τότε να αλλάξουν. Κάνω λόγο για την νομοθεσία, το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και για τα μέσα, τα αναγκαία κονδύλια, κονδύλια των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του εθνικού τομέα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Πιστεύω ότι πολλά χρήματα στοχεύουν στην κατάρτιση και εκπαίδευση των ανθρώπων, όμως δεν γίνονται όλα αυτά με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Απλά και μόνο κατάρτιση, κατάρτιση ε, προσφέρεται αλλά δεν προετοιμάζονται τα άτομα αυτά με τον καλύτερο τρόπο όπως θα έπρεπε. Κάτι άλλο που θα ήθελα να προσθέσω. Στη στρατηγική για το 2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί και στοχεύει η Ευρώπη να είναι η πιο ανταγωνιστική και η πιο προηγμένη περιοχή, ε, ήπειρος παγκόσμια δεν πρέπει να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια και να μείνουμε αδρανείς. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε να υπάρξουν αλλαγές, βαθιές αλλαγές και τομές. Αλλαγές για να αλλάξουν οι σημερινές τάσεις και οι σημερινές καταστάσεις. Πρέπει να αναθεωρήσουμε και να επανεξετάσουμε όλα. Το 2007 με, σε υπουργικό επίπεδο υπήρξε αναθεώρηση του εργασιακού κώδικα για τα θέματα τα οποία συζητούμε σήμερα. Στόχος ήταν να βελτιωθεί η δυνατότητα εργασίας ε, για τις γυναίκες και να συγκλίνει και να συμβιβαστεί και συνδυαστεί η επαγγελματική ζωή με την ε, οικογενειακή ζωή. Πέρασαν τέσσερα χρόνια από το 2007, σήμερα είμαστε στο 2011. Στον εργασιακό και οικογενειακό τομέα καλό είναι να θέλουμε να συνδυάσουμε τα πράγματα, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι πρέπει να υποπτεύουμε το τι γίνεται για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να εφαρμόζεται η νομοθεσία και όλοι να συμμορφώνονται για τους άνδρες και τους γυναίκες τις γυναίκες Σε ευχαριστούμε. Κύριε Αγουστίν, τώρα έχετε τον λόγο να απαντήσετε στις δύο αυτές ερωτήσεις που διατυπώθηκαν προηγούμενα από τον Μαλτέζο συνάδελφο και από την κυρία Μαζούρεκα της Πολωνικής Βουλής. Ευχαριστώ. Το πρώτο θέμα είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Όταν μιλάμε για δημογραφικά προβλήματα, εμείς δεν είμαστε τόσο αποπροσανατολισμένοι, δεν εργαζόμαστε μέσα σε ένα νομοθετικό κενό στο Βάγκουμ Legis. Υπάρχουν όμως πράγματα τα οποία έχουν αρνητικές επιπτώσεις. Και η αρνητική επίπτωση είναι η μεταφορά της εργασίας των θέσεων απασχόλησης προς προορισμούς όπου η εργασία στοιχίζει λιγότερο. Αλλά τη μετανάστευση αυτήν των επιχειρήσεων, μετατόπιση των επιχειρήσεων γίνεται και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτή την περίπτωση το πρόβλημα αφορά και τους νέους και τους γερούς. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν υπάρχει μία ενιαία συνταγή. Εγώ στην εισαγωγή μου προσπάθησα να πω ότι μπορούμε να κάνουμε εμείς Για παράδειγμα, μπορούμε να λύσουμε ορισμένα κοινωνικά ζητήματα, χωρίς όμως να ξεχάσουμε την αγορά, διότι η ενίσχυση του κοινωνικού συστήματος μπορεί να δημιουργήσει μια νέα αγορά. Στοιχίζει λιγότερο από τη συντήρηση των ανέργων ή η, βοήθεια, η βοήθεια εάν στο ιδιωτικό χρήμα προσθέσουμε και κρατικά κονδύλια από τον προϋπολογισμό όπως γίνεται στη Γερμανία θα έχουμε μία πλούσια αγορά παροχής υπηρεσιών με δημιουργία πολλών θέσεων απασχόλησης. Και μετά έχουμε το θέμα της συνεργατικότητας. Εμείς μάθαμε ότι θα πρέπει να οργανωθούμε και εμείς από μόνοι μας για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης. Εμείς ξεφορτώνουμε πάντα την ευθύνη στο κράτος ή στους εργοδότες. Αλλά όπως και η Ιταλία και η Πολωνία χρειάζεται μια αντίληψη κοινωνικής οικονομίας. είναι πολύ καλύτερο σε τοπικό επίπεδο οι άνεργοι να αυτοαπασχολούνται από ότι το να συνεχίσουμε εμείς να χορηγούμε επιδόματα ενεργείας. Το πρόβλημα της ε, παγκοσμιοποίησης δεν μπορεί να απαντηθεί παγκόσμια, πρέπει να έχουμε τοπικές απαντήσεις και το θέμα της, ε, των δυνατοτήτων των ηλικιωμένων από επαγγελματικής πλευράς το αγνοούμε πολλές φορές και έχουμε κατασπατάληση δυνάμεων. Πώς να χρησιμοποιήσουμε εμείς τους ηλικιωμένους ως εκπαιδευτές, ως ε, καθοδηγητές στην δουλειά των νέων στις επιχειρήσεις και με ευέλικτο ωράριο. Πολλές, ε, υπάρχουν μάλλον προγράμματα στην Ευρώπη που επιτρέπουν στους εργοδότες να χρησιμοποιούν ε, τις ε, δυνατότητες ε, αριστείας. Πώς μπορούμε όμως να το κάνουμε. Έχουμε εμεί τη γαλλική οργάνωση άκτη η οποία χρησιμοποιεί το δυναμικό της για να βοηθήσει όλους όσους αρχίζουν να φτιάχνουν τη δική τους επιχείρηση, να αυτοπασχολούνται, βοηθάνε τους νέους. Πρόκειται για μια ιδέα την οποία θα πρέπει να διαδώσουμε. Θα ήταν καλό αν αυτές ε, οι οργανώσεις ε, αυξανόντουσαν διότι οι ηλικιωμένοι αποτελούν ένα δυναμικό το οποίο θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Η συνάδελφος από την Πολωνία είπε κάτι με το οποίο συμφωνώ ότι οι γυναίκες είναι καταπληκτικές εργαζόμενες. Συχνά οι γυναίκες είναι αφοσιωμένες ε, στο χώρο εργασίας όσο και οι, γυναίκες, και άντρες. Ακριβώς επειδή υπόκεινται σε διακρίσεις, ε, δεσμεύονται τα διπλά, ε, προσπαθούν το διπλό για να μπορέσουν να πετύχουν και καλύτερα αποτελέσματα. Σίγουρα υπάρχει διάκριση κατά των γυναικών. Θα πρέπει να την καταπολεμήσουμε σίγουρα διαμφισβήτητα όλοι θα πρέπει να είμαστε από την ίδια μεριά του οδοφράγματος. Και με ευχαρίστησε και ένα άλλο σχόλιο. Για τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία υποχρησιμοποιούνται μα γι' αυτό το θέμα θα μπορούσε κανείς να γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο σε διάφορες χώρες και στη δική μου αλλά το, στην ουσία το ζήτημα δεν αφορά στη σπατάλη αλλά στην αποτελεσματικότητα αυτών των χρηματοδοτήσεων και αυτό διαφέρει σε, σε πολλά εμείς ε, στα κράτη-μέλη πρέπει να ξαναδούμε αυτά τα προγράμματα, να επιλέξουμε τα πιο αποτελεσματικά και να προχωρήσουμε. Διότι πολλά χρήματα τα οποία τα μοιράζουμε και τα ξαναμοιράζουμε σε σχέδια με μικρή αποτελεσματικότητα δεν χρησιμοποιούνται σωστά. και στο όνομα της πειθαρχία θα πρέπει να εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Πάντως, μην ξεχνάτε ότι ορισμένες πρωτοβουλίες θα πρέπει να τις εγκαταλείψουμε για να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στις γύρω τα πιο σοβαρά σχέδια και να κάνουμε ένα βήμα προς τα μπρος για το θέμα του monitoring όταν κοιτάμε εμείς τις δαπάνες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου υπάρχει πάντοτε ο τίτλος αξιολόγηση αλλά τι γίνεται μετά συμβαίνει κάτι όχι δεν συμβαίνει κάτι, κάτι το ιδιαίτερο δυστυχώς το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης πολλές φορές δεν αντικα τοπτρίζονται με τροποποίηση στα διάφορα προγράμματα ή με την επιλογή καλύτερων προγραμμάτων. Δεν φτάνει μόνο να αξιολογούμε, πρέπει να διδασκόμαστε κιόλας από αυτήν την αξιολόγηση. Υποστηρίζω ότι νέε προτάσεις κανονισμού, από όσα ξέρουμε γιατί ακόμη συζητιέται το πράγμα, θα διευκολύνουν την επιλογή μιας προσέγγισης που θα στοχεύει στην αποτελεσματικότητα. Χαίρομαι που έχουμε αυτή την απήχηση και από τα ε, εθνικά κοινοβούλια και όχι μόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ τον γερουσιαστή. Αυτό κλείνει τη συζήτηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ήθελα να ζητήσω από τον γερουσιαστή Αουγκουστίν αν θέλει να κλείσει τη συζήτηση. ή αν θεωρεί ότι ό,τι ήταν να ακουστεί έχει ακουστεί μέχρι τώρα. Ε, λέει ο ένα πράγμα να πω μόνο, το οποίο ίσως ξέχασα να αναφέρω προηγουμένως. Ο Στεφάν Κισινέσκι, ένας γνωστός δημοσιογράφος από την εφημερίδα της ε, Αλληλεγγύης, βλέποντας τα καθεστώτα τα, της Ανατολικής Ευρώπης που έπεφταν το ένα μετά το άλλο, είπε ότι δεν είναι η κρίση αυτή, είναι το αποτέλεσμα της κρίσης αυτό που βλέπουμε. Και η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίση, αλλά δεν είναι σε κρίση πραγματικά, είναι στο αποτέλεσμα της κρίσης και μιας τεράστιας έλλειψης δράσεων μιας μεγάλης αδράνειας. Το θέμα δεν είναι να κόβουμε λεφτά δεξιά και αριστερά. Προφανώς πρέπει να είμαστε επιθαρχημένοι, αλλά πρέπει να είμαστε λογικοί, να μην ξεχνάμε την αρχή της αλληλεγγύης και να προσπαθήσουμε στο μέλλον να προλάβουμε τέτοιες καταστάσεις και να καλυφθούμε, γιατί η Ευρώπη είναι σαφές ότι καθυστέρησε και αντέδρασε σε κάποια προβλήματα τα οποία τέθηκαν και δεν προσπάθησε να τα προβλέψει. Ελπίζω λοιπόν το νέο αυτό πακέτο να δώσει μια νέα θα έλεγα προοπτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να λειτουργήσει επιτέλους προληπτικά και όχι να περιμένει διορθωτικά να ανακάμψει. Αυτό. Τίποτα περισσότερο πρόεδρο. Ευχαριστώ κύριε Αγκουστίν. Αυτό κλείνει τη συζήτησή μας σε αυτό το τρίτο πάνελ. Θα περάσουμε τώρα στην Ολομέλεια σε λίγα λεπτά. Θα προεδρεύσει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Γεύζη Μπούζεκ. Πέντε λεπτά διάλειμμα. Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε στα έδρανά σας. Θα ξεκινήσουμε αμέσως με τη συνεδρίασή μας. Αυτή της τελευταίας ολομέλειας πριν από το τέλος και ολοκλήρωση της ε, συνεδρίασής μας, της κοινή κοινοβουλευτικής συνεδρίασής μας. Και θα ολοκληρώσουμε έτσι με την τελευταία μας ολομέλεια. Απλώς ανοίγω αυτή την ολομέλεια στις εργασίες της και πάλι. Θα είναι ένας γύρος, μια ολομέλεια που θα αφιερωθεί στον κύριο ε, Βραντίσλαφ Κόντζες που είναι υπεύθυνος ε, εκπρόσωπος ε, της Πολωνικής Προεδρίας και του κυρίου Λάσλο Άντορ Επιτρόπου για την απασχόληση κοινωνικές ε, υποθέσεις ε, και κοινωνική ένταξη και ολοκλήρωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μετά από αυτές τις παρεμβάσεις θα διεξαχθεί συζήτηση. Αν θέλετε να συμμετάσχετε σε αυτή τη συζήτηση, παρακαλώ να συμπληρώσετε τα έντυπα τα, ε, της αίτησης, του αιτήματο για παρέμβαση στην Ολομέλεια. Οι κλητήρε, οι κλητήρες που είναι παρόντες εδώ στην αίθουσα θα σας δώσουν θα δοθεί ε, αυτή η ε, αίτηση ε, και σε λίγα λεπτά θα μπορέσει να διατεθεί αυτή, να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα μπορείτε να έχετε τα έντυπα, τα οποία όταν θα τα συμπληρώσετε θα τα παραδίδετε πάλι στους ίδιους κλητήρες για να φτάσουν ως εμάς. Και μετά θα ξεκινήσουμε με τις παρεμβάσεις στη συζήτηση. Πρώτα θα έχουμε δύο παρεμβάσεις, εισαγωγικές παρατηρήσεις του κυρίου Βλαντίσλαβ Πόσνια και του κύριου Επιτρόπου Άντορ. Αυτές τις δύο ε, εισηγήσει θα ακούσουμε πρώτα. Και μετά θα έχουμε τρεις, ε, τριών λεπτών παρεμβάσεις. Θα προετοιμαστεί ο πίνακας, ο κατάλογος των αγοριτών που θα παρέμβουν με βάση τα έντυπα, τα, τα έντυπα των αιτήσεων που θα έχετε συμπληρώσει για τις παρεμβάσεις σας θα προετοιμαστεί, θα καταρτιστεί αυτός ο πίνακας αγοριτών και έχουμε επίσης και τη σειρά μας, θα έχουμε και την εξή σειρά παρεμβάσεων. Δύο εκπρόσωποι εθνικών κοινοβουλίων, ένας ευρωβουλευτής και πάλι εναλλάξα δύο ε, εκπρόσωποι εθνικών κοινοβουλίων, ένας ευρωβουλευτής και ούτω καθεξής. Τρία λεπτά για κάθε παρεμβαίνοντα για κάθε αγορητή. Και κάτι άλλο το οποίο είναι και αυτό σημαντικό. Αν θέλετε να ρωτήσετε, να θέσετε μία ερώτηση ή να κάνετε κάποιο σύντομο σχόλιο σε κάποιον προλαλήσαντα αγορητή, μπορείτε να σηκώσετε την μπλε κάρτα. Εγώ ελπίζω ότι έχετε αυτές τις μπλε κάρτες. Εγώ δεν έχω κάποια τέτοια μπλε κάρτα να σας την δείξω. Μια μπλε κάρτα, κιανή κάρτα. Αυτό μόνο σε περίπτωση που θέλετε να διατυπώσετε ένα ερώτημα ή να κάνετε ένα σύντομο σχόλιο. Και μετά μπορεί να υπάρξει σύντομη απάντηση. 20 δευτερόλεπτων, μισού λεπτού το πολύ απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις ή σχόλια. Επιπρόσθετα στον χρόνο αγόρησης που θα έχετε, αν έχετε εγγραφεί στον κατάλογο αγορητών. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δυνατότητα. Όλα λοιπόν νομίζω είναι πλέον απόλυτα σαφή. Θα μπορούσαμε άμεσα να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Θα ήθελα με ιδιαίτερη χαρά να σας δώσω τον λόγο, κύριε Κάμισε που εκπροσωπείται την κυβέρνηση ακριβώς της Πολωνίας και την Πολωνική Προεδρία του Συμβουλίου. Θα ήθελα, όπως σας ανέφερα, να κάνετε αυτή την εισαγωγή, την ε, εισαγωγική εισήγησή σας και έτσι μετά να ξεκινήσουμε και αργότερα τη συζήτηση. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε και εσάς, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Εξ ονόματος του Πρωθυπουργού της Πολωνίας, κυρίου Ντόναλντ Τούσκ, εξ ονόματος της Πολωνικής Προεδρίας σας ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση να συμμετάσχουμε στη σημερινή συζήτηση και για την δυνατότητα που μας προσφέρετε να παρουσιάσω σήμερα τις θέσεις της Πολωνικής Προεδρίας για τόσο σημαντικά θέματα όπως τις δημογραφικές εξελίξεις και την κοινωνική πολιτική. Είναι τιμή και είναι πραγματικά μια ευκαιρία για να ακούσω και τις δικές σας απόψεις όσον αφορά τη διάγνωση που γίνεται για αυτή την κατάσταση και τις προτάσεις σας. Κυρίες και κύριοι, τον 20ο αιώνα, ο 20ος αιώνας ήταν ένας αιώνας μιας έκρηξης στον τομέα της υγείας. Είδαμε πως πολλαπλασιάστηκε, τέτραπλασιάστηκε κιόλας ο παγκόσμιος πληθυσμός μέχρι τα 6 δισεκατομμύρια ε, κατά τα τέλη του 2000. Ε, και πρόσφατα είδαμε πώς γεννήθηκε, ότι γεννήθηκε και ε, ολοκληρώθηκε το 7ο δισεκατομμύριο από πλευράς παγκόσμιου πληθυσμού. Θα είναι όμως αυτός ο αιώνας, ο 21ος αιώνας, μια προοπτική με φθήνουσα, με φθήνον πρόσημο ε, μείωσης και συρρήκνωσης για τον πληθυσμό της Ευρώπης δημογραφικά. Στην Ευρώπη έχουμε μια ιδιομορφία. Αυτή η ιδιομορφία είναι η εξής. Πρώτα, είδαμε τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής της κατάστασης και είναι αναγκαίο να υπάρξει ένας πόλος ε, ενδυνάμωσης ε, και αλλαγής. Πολλοί επαΐοντες λέγουν ότι συμφωνούν για το ότι μια κοινωνία όλο και περισσότερο ηλικιωμένων ανθρώπων που γυράσκει όλο και περισσότερο θα έχει τη συνιστόσα των μεταναστών σε, ως τμήμα αυτής της κοινωνίας. Αλλάζει λοιπόν η κοινωνία, το βλέπουμε στην ευρωπαϊκή κοινωνία σήμερα. Και αν θέλουμε στον επόμενο αιώνα να υλοποιηθούν αυτές οι προοπτικές, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα του συρρυκνούμενου πληθυσμού και του μικρότερου ε, ποσοστού στον παγκόσμιο πληθυσμό από πλευράς της Ευρώπης. Έχουμε πολλές μελέτες και πολλές ε, ε, τοποθετήσεις δεν είναι μόνο κάτι ε, φυσικό ή ένας φυσικός νόμος ή απομάκρυνση από τις ε, ε, επαγγελματικές δραστηριότητες, δηλαδή η συνταξιοδότηση και η αποχώρηση από τον επαγγελματικό βίο. Καθόλου φυσικό δεν είναι αυτό, είναι απλώς κάτι το οποίο απορρέει από νομοθεσίες. Υπάρχει και ένα δαπανηρό πλαίσιο και πέρα από το ε, νομικό πλαίσιο που ξεπερνά αυτή η κατάσταση το νομικό πλαίσιο. Το πρόβλημα που έχουμε επιπλέον είναι η κρίση, η δημοσιονομική και χρηματοοικονομική κρίση και γι' αυτό πρέπει να εξισορροπηθούν οι προϋπολογισμοί. Είναι πολύ εύκολο να κάνουμε λόγο για κοινωνικά θέματα σε μια περίοδο κοινωνικής οικονομικής Είναι πολύ πιο δύσκολο όμω να γίνεται λόγος για τέτοια πράγματα σε μια περίοδο κρίσης. Έχοντα ε, αναφέρει αυτά τα πράγματα σε σχέση με την ε, ε, λιδία λίθο που έχουμε τώρα για να δούμε αν θα είμαστε ικανοί να είναι αξιόπιστο το ευρωπαϊκό πρότυπο και να είναι βιώσιμο. Ακριβώς τώρα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. Αποφάσεις που μπορούν να ενδυναμώσουν την ανταγωνιστικότητα από πλευρά της Ευρώπης και να ενδυναμώσουν και να τονώσουν την ε, κοινωνική και οικονομική συνοχή της Ευρώπης. Γι' αυτό είναι σκόπιμο το δημογραφικό πρόβλημα και τα θέματα τα κοινωνικά να εγγραφούν, να έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη αυτής της συνάντησης εθνικών βουλευτών και ευρωβουλευτών για την εξέταση αυτών των ζητημάτων. Και επιπλέον θα ληφθούν και αποφάσεις μέσα σε αυτά τα πλαίσια από εσάς για τις τελικές λύσεις που θα υιοθετηθούν. Κυρίες και κύριοι, η ανάλυση των σημερινών δημογραφικών τάσεων καταδεικνύει ότι ο πλούτος των πολιτών και ένα υψηλό επίπεδο, η ευημερία και ένα υψηλό επίπεδο κοινωνικής ασφάλισης ε, δεν είναι σε μια περίοδο κρίσης ο εχθρός ε, του να αποκτά κανείς παιδιά. Πρέπει να βρούμε πολιτικές και μέσα για να υποστηρίξουμε τις οικογένειες, να συγκλίνει και να συνδυαστεί η επαγγελματική ζωή με την οικογενειακή ζωή, να επιτευχθεί ισότητα στον εργασιακό τομέα, στην εργασία αλλά και στην οικογένεια μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και πέρα από αυτό είναι αναγκαίο να επενδύσουμε στην παιδεία, εκπαίδευση και κατάρτιση και στην επιμόρφωση και στην επαγγελματική κατάρτιση και ιδιαίτερα όσον αφορά και τους ε, ηλικιωμένους. Οι δημογραφικές αλλαγές στην Ευρώπη όχι μόνο απαιτούν να υπάρξει μεγαλύτερη καινοτομία στις δράσεις μας, αλλά πρέπει να διευρύνουμε τις πολιτικές και τις ε, δυνατότητες ε, που διατίθενται για την επίτευξη των στόχων. Αυτό πρέπει να γίνει. Η εργασιακή αγορά εργασίας απαιτεί να υπάρχει συμμετοχή των γυναικών στο επαγγελματικό επαγγελματικό τομέα. Και πρέπει και νέοι επίσης να μπορούν να απασχοληθούν. Είναι σημαντικότατοι αυτή η στόχη και πρέπει να προωθηθεί η συμφιλίωση, η σύγκληση των οικογενειακών με τις επαγγελματικές δραστηριότητες και να μπορέσουν να επιμεριστούν, ε, να κατανεμηθούν οι υποχρεώσεις ε, επαγγελματικές και οικογενειακές μεταξύ ανδρών και γυναικών με ίσο, ίδιο, ισοδίκιο τρόπο. Πρέπει να είναι δυνατή η απασχόληση και η προώθηση της απασχόλησης στην ηλικία 50 συν. Θα πρέπει να δούμε πολύ ε, πιο ισχυρή συμμετοχή, μια και αυτή θα αντιπροσωπεύει αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μεγαλύτερο ε, τμήμα της κοινωνίας ε, μέσα από τη διαδικασία υπεργύρασης. Ε, είναι μια γενεά που είχε μια πολύ και έχει μια πολύ καλή επαγγελματική κατάρτιση και έχει τύχει πολύ καλής παιδείας. Η συμμετοχή αυτών των ατόμων στην κοινωνία μας είναι ένας πλούτος στην, για την κοινωνία της Ευρώπης όσον αφορά την επόμενη δεκαετία και το μέλλον. Αναφέρθηκε πιο πριν πέρα από τα δημογραφικά προβλήματα της Ευρώπης πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη ότι αυτό θα πρέπει να είναι και ένα από τα κέρια σημεία δράσης ε, του Συμβουλίου. Κάνουμε λόγο για τη δημογραφία, δημογραφικά θέματα, για το μέλλον της Ευρώπης. Ε, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εθελοντικής ε, συμμετοχής και απασχόλησης και δράσης πρέπει δίνοντας συνέχεια σε αυτά τα οποία κάνουμε, δίνουμε συνέχεια στις προηγούμενες προεδρίες και δράσεις τους, όπως της Γερμανικής προεδρία, να πάρει ευρωπαϊκή διάσταση αυτό το θέμα, αλλά και η Τσεχική, η Ουγγρική, η Σουηδική και άλλες προεδρίες έχουν ακριβώς επικεντρωθεί σε αυτά τα θέματα των δημογραφικών προβλημάτων. Εγκρίθηκαν από πλευρά Συμβουλίου μια σειρά συμπερασμάτων για μια καλύτερη διευρυμένη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργανών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμβουλίου, Επιτροπή Ευρωκοινοβουλίου για την κοινωνική πολιτική, την πολιτική απασχόληση και για την οικονομική πολιτική Καλύτερε δυνατότητε συντονισμού και δράσεων. Αυτό θα επιτρέψει να υπάρξει μια ανταλλαγή, μια πιο συστημική και συστηματική ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, βέλτιστων πρακτικών. Με αυτόν τον τρόπο να προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσει στι προκλήσει ε, τι δημογραφικέ που αντιμετωπίζουμε αντιμετωπίζουμε ώστε να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε και να πετύχουμε τους στόχους μας. Με αυτές ε, τις πρωτοβουλίες και στόχους η Πολωνική Προεδρία οδήγησε στο να εγκριθεί από το Συμβούλιο μια σειρά συμπερασμάτων για την ε, υπεργύρανση του πληθυσμού της Ευρώπης ε, και το συσχετισμό αυτών των θεμάτων με την αγορά εργασίας. Συνδυασμό δηλαδή δυνατοτήτων που θα δίνει δυνατότητα να επιλεγούν οι θετικές πτυχές δράσης. Η οικονομία που θα συμπεριλαμβάνει τους ηλικιωμένους αλλά και θα δίνει και ευκαιρίες στους νέους. Κυρίες και κύριοι, η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 πρέπει να επιτύχει την ε, ανάπτυξη και θα είναι η λιδία λίθος ε, αυτή για την επίτευξη των στόχων μας. Πολλές φορές η υπεργύρανση, η ύπαρξη όλο και περισσότερων ηλικιωμένων αφορά και δημιουργεί πίεση όλο και μεγαλύτερη για να γίνει κάτι ε, ε, σε αυτό το πεδίο. Οι δημογραφικές αλλαγές κυρίες και κύριοι μην ε, εξελίσσονται μπροστά μας, μπροστά στα μάτια μας και είμαστε παρατηρητές τους. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση δεδομένης της επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Δεν υπάρχει χρόνος να σπαταληθεί. Πρέπει να συνδυαστεί η επαγγελματική ζωή με την ε, οικογενειακή ζωή. Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή. Είναι ύψιστη η σημασία αυτής της αξίας και αρχής. Είναι αρχές και αξίες που μας ενώνουν πανευρωπαϊκά αυτές. Κυρίες και κύριοι, να σωθεί η Ευρώπη από την κρίση. Δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί η Ευρώπη και δεν πρέπει να σταυρώσουμε τα χέρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσίασή σας. Όλα τα σχόλια. Και συνεχίζει στα αγγλικά. Και τώρα θα λάβει τον λόγο ο κύριος Λάσλο Άντορ, επίτροπος. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, Πρόεδρε, βουλευτές, ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, είναι χαρά για μένα να βρίσκομαι εδώ για να συζητήσουμε θέματα που έχουν τόσο σήμαν μεγάλη σπουδαιότητα για την κοινωνία μας και το μέλλον των κοινωνιών μας, κοινωνική συνοχή και δημογραφικές αλλαγές. Αυτά τα θέματα είναι ακόμα πιο σημαντικά σήμερα στην σημερινή χρηματοοικονομική νομισματική κρίση που περνάμε. Η ευρωπαϊκή δημογραφία αλλάζει. Ο πληθυσμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση γυράσκει. Η γεννητικότητα, ξέρετε ότι σε πάρα πολλές χώρες έχει ξεκινήσει μια μειωτική τάση και ακόμα και ο απόλυτος αριθμός του πληθυσμού ε, φαίνεται ότι θα μειωθεί στο μέλλον. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας δυσκολίες. Ήδη από τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε μια ανακοίνωση σε σχέση με τις πολιτικές απαντήσεις στην δημογραφική κρίση. Η τελευταία όμως οικονομική κρίση είναι κάτι το οποίο περιορίζει τις δυνατότητες κίνησης που έχουμε στον τομέα αυτό. Για να μπορέσει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει θα πρέπει παρά τις δυσκολίες τις οποίες συναντάμε να προσπαθήσουμε να πετύχουμε τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει στα πλαίσια της Ευρώπης του 2020 γιατί η ευημερία της Ευρώπης δεν εξαρτώνται μόνο από την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα, αλλά και από την ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου, των ανθρώπινων πόρων και την κοινωνική συνοχή. Η επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξαρτηθεί κατά πολύ και από την απάντηση που θα δώσουμε στις δημογραφικές απειλές. Βασικά χαρακτηριστικά της στρατηγικής αυτής είναι πρώτον να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα ποσοστό ανεργία το οποίο να θεωρείται ανοιχτό, να είναι χαμηλότερο εν πάση περιπτώσει από το σημερινό και να μειώσουμε και τον αριθμό των λεγόμενων πτωχών από το 2015 και μετά. Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να διευρύνουμε τη συνεργασία ανάμεσα στις διαφορετικές γενναίες και να δώσουμε περισσότερες δυνατότητες στους ηλικιωμένους. 45% ε, των, εργαζομένων ήσαν κάτω το 64, των 64 ετών. Θα πρέπει αυτό δεν αρκεί να μεγαλώσει το ποσοστό ακόμα περισσότερο. Οι εργαζόμενοι άνω των 50-60 ετών είναι διαθέσιμη και πρέπει να είναι διαθέσιμη για την αγορά εργασίας. Ε, ξέρετε ότι πολλοί κόσμος σταματά την επαγγελματική του δραστηριότητα ενωρίτερα των 65 ετών και μάλιστα η μέση όρη σε πάρα πολλές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν είναι άνω του 61 και 62 ετών. Πιστεύουμε ότι τα δημοσιονομικά θα πρέπει να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση και θα πρέπει να μας επιτρέψουν να περιορίσουμε την πρόορη συνταξιοδότηση και να προβλέψουμε και μια παράταση της επαγγελματικής δραστηριοποίησης η οποία να συμβαδίζει με την παράταση της ε, επιβιωσιμότητας των πολετών. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να επωφεληθούμε από την ε, μεγαλύτερη διάρκεια της ε, ε, ζωής των πολιτών σήμερα και να υπάρξει μια αντίστοιχη αύξηση και της επαγγελματική τους δραστηριότητας χρονικά ενώ. Οι πολίτες οι οποίοι συνταξιοδοτούνται σε μια κάποια ηλικία πρέπει να νιώθουν χρήσιμοι Πρέπει να νιώθουν χρήσιμοι ανεξαρτήτως της ηλικίας τους. Πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε ειδικά μέτρα για τους ηλικιωμένους εργαζομένους. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε και να ανοίξουμε τις δυνατότητες τους ηλικιωμένους έτσι ώστε να καταστούν ελκυστικοί για την αγορά εργασίας. Νομίζω ότι αυτό θα είναι εγγύηση για μια ευρυθμότερη λειτουργία της κοινωνίας μας για όλες τις ηλικίε. Ήδη από τον επόμενο χρόνο θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για την προώθηση όλων αυτών των ιδεών μέσω ενός σχεδίου, ενός προγράμματος διαγενειακής αλληλεγγύης. Το 2020, το 2012, συγγνώμη, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις προϋποθέσεις που θα διασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για τους νέους αλλά και για τα ηλικιωμένα μέλη της κοινωνίας μας. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με προσεκτικό τρόπο είναι οι ανισότητες στην Ευρώπη. Βλέπουμε πάρα πολλά δείγματα αυτών των ανισοτήτων στην Ευρώπη. Πάρα πολλοί πολίτες έχουν απογοητευτεί από την πολιτική, από την οικονομία και από την κοινωνία. Η αλωτρίωση των πολιτών ε, είναι κάτι το οποίο υπονομεύει το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο, υπονομεύει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και φυσικά υπονομεύει και την έξυπνη και διαρκή ανάπτυξη. Δεν μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους αυτούς αν δεν σταθούμε πιο συμπεριληπτικοί ενώ σε επίπεδο πληθυσμών στα πλαίσια της προσπάθειας για ανάπτυξη. Υπάρχουν προβλήματα ανισοτήτων, υπάρχουν προβλήματα ανισοτήτων σε γεωγραφικό επίπεδο, σε επίπεδο χωρών, και να δούμε λίγο καλύτερα και τον ρόλο των περιοχών που βρίσκονται σε ε, μεγάλη απόσταση από τα κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανισότητες σε επίπεδο εισοδημάτων των κατοίκων των διαφόρων περιοχών έχουν ε, λίγο μειωθεί, αλλά παρόλα αυτά η κατεύθυνση θα πρέπει αυτή να συνεχιστεί. η σωστή εφαρμογή των διαθέσιμων πολιτικών μέσων θα μπορέσει να μας βοηθήσει να επηρεάσουμε θετικά τις δημογραφικές εξελίξεις. Και δεν θα πρέπει να βλέπουμε τις δημογραφικές εξελίξεις σαν ένα πρόβλημα, αλλά σαν μια ευκαιρία, σαν μια δυνατότητα. Το πρόβλημα βέβαια το οποίο τίθεται με πάρα πολύ οξύ τρόπο σήμερα είναι η ανεργία των νέων. Οι νέοι έχουν δύσκολη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν χιλιάδες επιχειρήσεις οι οποίες προσπαθούν να αναζητήσουν και να βρουν το κατάλληλο και το σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό. Υπάρχει μια έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού που θα βοηθήσει σε αρνητικά το λέω αυτό να καταλήξουμε σε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης στην Ευρώπη. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε είναι το θέμα της μετανάστευσης θα πρέπει να υπάρξει μια μεταναστευτική πολιτική με βάση τις ικανότητες στην εργασία των μεταναστών. Θα πρέπει επίσης να εναρμονίσουμε και τα συστήματα κοινωνικής κάλυψης, όπως επίσης και τα συστήματα αναγνώρισης ε, των διπλωμάτων και των ικανοτήτων των εργαζομένων για να διευκολύνουμε την ε, κινητικότητά τους. Έτσι μόνο η πολιτική της μετανάστευσης θα επιτρέψει και στους μετανάστες να έχουν σωστή πρόσβαση στην αγορά απασχόλησης. Μέσω του προγράμματος Ευρώπη 2020 θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε την συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης κοινωνικά και εδαφικά, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα τα οποία θέτει στη διάθεσή τους η Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι να τερματίσουμε τις διαφορές ανάμεσα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι μόνο θα προστατεύσουμε τις πιο ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού έτσι θα προχωρήσουμε σε δημοσιονομική εξυγίανση και θα μπορέσουμε ε, να ξεφύγουμε από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει από τα κράτη-μέλη να ε, μην κλονίσουν τον σταθεροποιητικό ρόλο της κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής κάλυψης. Αυτό σημαίνει ότι οι πολιτικές μας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο χρήζουν περαιτέρω συντονισμού και συνεργασία στο σχεδιασμό τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα ξεκινήσει η συζήτηση. Πρώτος ομιλητής, ο εκπρόσωπος του Πορτογαλικού Κοινοβουλίου, Νούνιο Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα θέλω να χαιρετήσω αυτή την πρωτοβουλία για τη στιγμή στην οποία διαδραματίζεται και συμβαίνει, αλλά επίσης και για το θέμα που έχουμε τη συνειδητοποίηση και το θάρρος να εγγράψουμε στην κοινοτική μερίσια διάταξη. Και δεύτερο, να τονίσω ότι αυτές οι συναντήσεις αντανακλούν και ενισχύουν ένα πνεύμα αλληλεγγύης Κοινοτική αλληλεγγύη που μας βοηθά να υλοποιήσουμε και να εξειδικεύσουμε το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Είμαστε εδώ επειδή ο χρόνος και η στιγμή προβληματισμού απαιτούν δράση, απαιτούν απαντήσεις σε αξίες πολιτισμικές που αναπτύχθηκαν και υλοποιήθηκαν από την Ευρώπη και που ήταν και είναι σημαντικά στοιχεία για την διατήρηση και την αηφορία τους χωρίς να υπονομεύεται με κανένα τρόπο η δυνατότητα δημιουργίας, καινοτομία και ενδυνάμωσης και τόνωσης των αξιών και αρχών μας. Διότι αυτό, αυτό είναι το κύριο σημείο της παρέμβασής μου. Η Ευρώπη από πλευρά της ιστορίας της ήταν φάρος, παγκόσμιος φάρος για το υπόδειγμα, το πρότυπο των αρχών, των αξιών, της πολιτισμικής δράσης αλλά και της αηφορίας και της μορφής αηφορίας για αυτά τα κεκτημένα. Αυτός ήταν ο πλούτος που υπήρχε και είχε η Ευρώπη για να διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα και που έπρεπε να διατηρηθεί. Αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Η Ευρώπη μέσα στο πλαίσιο μια παγκοσμιοποιημένη, όλο και πιο ανοιχτή οικονομία που λιγότερο αναπτύχθηκε σε σχέση με άλλε οικονομικέ μονάδε άλλων υπήρων πρέπει να διασφαλίσει την ανάπτυξή τη ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί την αηφορία τη αυτών των πολιτισμικών αρχών και αξιών που είμαστε δημιουργοί στο παρελθόν. Και γι' αυτό σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσουμε ότι είναι πρωταρχική σημασίας να μην αγνοήσουμε αυτό τον πλούτο που μπορούμε να δημιουργήσουμε και που μπορούμε να υλοποιήσουμε όπως και που πολλές φορές δεν ε, επιτυγχάνεται και το, όπως απαιτεί και το κοινωνικό ευρωπαϊκό πρότυπο που πρέπει να διασφαλιστεί. Αυτή τη στιγμή συνειδητοποιούμε ότι και αυτές οι ατέλειες και ελλείψεις στον οικονομικό τομέα δημιούργησαν ένα σύνολο οικονομικών συντελεστών και στοιχείων αλλά και δημογραφικών που υπονομεύουν την αηφορία. Πρέπει όμως ανυποχώρητα να συντηρήσουμε και να διασφαλίσουμε το ευρωπαϊκό πρότυπο, κοινωνικό ευρωπαϊκό πρότυπο. Πρέπει να βρούμε τις απαντήσεις που χρειαζόμαστε και να μην τις ξεχάσουμε ούτε μια στιγμή και να μην καθυστερήσουμε καθόλου. Πρώτον, πρέπει οι πολιτικοί ηγέτες να επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στις επόμενες γενναίες και λιγότερο στι μελλοντικέ εκλογικέ αντιπαραθέσει. Οι πολιτικές στην κοινότητα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχουν την ελαστικότητα και ενδυνάμωση μέσω μέσων και κονδυλίων που θα μπορούν να διασφαλίσουν τις πολιτικές και οικονομικές δράσεις για την οικονομική ανάπτυξη. Και ένας τρίτος άξονας σημαντικός θα πρέπει να δοθεί με σημαντική προσοχή στο ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο. Αυτή την κοινωνική Ευρώπη που πρέπει πέρα από τις γενναίες να διασφαλίσουμε. Τέταρτο σημαντικό στοιχείο Πάλι εμεί, οι Ευρωπαίοι και όλα τα τμήματα αυτή της μεγάλης Ευρώπης να βοηθήσουμε όλοι αυτές οι πολιτιστικές αξίες να να διαχέονται παγκόσμια, να μπορούν να διαδίδονται παγκόσμια, να μην υπάρξουν στρεβλώσεις όσον αφορά την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας που σήμερα δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες και δημιουργεί οι προϋποθέσεις που δεν συνεισφέρουν στην αηφορία. Πιστεύουμε ότι αυτές οι συζητήσεις είναι πολύ σημαντικές. Βοηθούν να καταλάβουμε και να αντιληφθούμε ότι υπάρχει ένα σύνολο θεμάτων για την ε, ανάπτυξη που πρέπει να προσέξουμε ώστε να είμαστε κοινωνικά και πολιτισμικά όπως πάντα είμαστε ένα πρότυπο για τον πολιτισμένο κόσμο. Ευχαριστώ. E, Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ συνάδελφε, εκπρόσωπος της Γαλλικής Γερουσίας, ο Ζων Λουί Λογά. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, οι χθεσινές και σημερινές μας συνεδριάσεις που αφιερώσαμε στις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της δημογραφικής εξέλιξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα εν μέρει αρνητικό. Όχι, όχι οι εργασίες μας, αλλά η διαπίστωση. Δηλαδή, εμείς ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι διαπιστώνουμε, βλέπουμε τα κράτη μας να υπόκεινται τις ε, ε στρεβλές επιπτώσεις ε, της ε, παγκοσμιοποίησης, να υπόκειται την κρίση και βλέπουμε να ξαναζωντανεύει η μια φτώχεια που την είχαμε ξεχάσει από το 1945 και μετά φτώχεια η οποία θα πλήξει ακόμη και τα παιδιά. Η φιλοδοξία των πατέρων ιδρυτών της Ένωσης ήταν η πρόοδος και η ευημερία. Η πρόοδος μέσα στην ευημερία. Εμείς διαπιστώνουμε ότι έχουμε μεταναστευτικούς πληθυσμούς. Όχι μόνο αυτούς που πρέπει εμείς να υποδεχθούμε και όχι με οποιονδήποτε τρόπο που αποτελούν ελπίδα κατά της γύρανσης του πληθυσμού μας και που λόγω προκαταλήψεων εμείς θέλουμε να τους στείλουμε από πίσω, πίσω εκεί που μας ήρθαν. Βλέπουμε λοιπόν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες ε, οι πολίτες ε, κυρίως για τα θέματα πρόσβασης ε, στον τομέα της υγείας. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να, κατεβα... να... να κατεβάσει τα χέρια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ ως γιατρός είμαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος στο θέμα της πρόσβασης ε, στις ε, θεραπείες και στις φροντίδες. Θα έπρεπε να φροντίσουμε να έχουμε εναρμόνιση των πτυχίων στον ε, τομέα της υγείας για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε επίσης και τη διασυνοριακή συνεργασία και να εξορκίσουμε τον κίνδυνο της έλλειψης ιατρών. Επίσης υπάρχει το θέμα των καθολικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος. Και ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να θέλω να είμαι εθνικιστής, έχει πρόβλημα γύρω από αυτό με τον Επίτροπό μας, τον κύριο Μπαρνιέρ. Η Ευρώπη για μας δεν είναι μόνο μία αγορά το γεγονός ότι αμφισβητείται σήμερα λόγω της ε, κρίσης ε, θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αποκαθιστώντας τον κοινωνικό τομέα και προστατεύοντας τον πολίτη που θα μπορούσε αυτό να αποκαταστήσει και τη φήμη της. Εμείς ε, στην Γερουσία έχουμε μια πραγματική συζήτηση για τις αξίες μέσα στη δράση που καθορίζονται από την ηθική ηθική που θα πρέπει να αναπτύξουμε και στην Ευρώπη τόσο στον τομέα της ε, κατάρτισης όσο και της έρευνας. Ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτησή σας, λέει ο κύριος Μπούσεκ. Δίνω το ε, δίνω τώρα την, το λόγο στον κύριο Μπουρόσεβιτς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και στη, για την κυρία Γιαζοβιέσκα θα λάβετε τον λόγο από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ. Ο κύριος Επίτροπος ε, στον λόγο που εξεφώνησε τόνισε ότι Μία από τις αρχές και αξίες της επιτυχίας της Ευρώπης μπορεί να είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Κύριε Πίτροπε, πιστεύω απόλυτα αυτό το πράγμα. Είναι η ανώτατη αξία το ανθρώπινο δυναμικό που έχει η Ευρώπη στη διάθεσή της. Φανταστείτε έναν κόσμο ο κόσμος που αλλάζει από τους Ευρωπαίους, από τους Ευρωπαίους και οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Κίνα για παράδειγμα με τις πολλές εταιρείες που έχουν σίγουρα όμως το ταλέντο, το ανθρώπινο δυναμικό και οι ικανότητες. Η καινοτομία και οι νέοι τρόποι σκέψης ε, είναι κάτι που έχει η Ευρώπη ως δυναμικό στα χέρια της. Είναι ένα μήνυμα, ένα χαρτί, ένα ε, δυναμικό ε, που πρέπει να χρησιμοποιήσει ως δυνατό χαρτί η Ευρώπη παγκόσμια. Κάνουμε λόγο για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με ησυχάζει το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τα κονδύλια του θα χρησιμοποιούνται για την ε, ε, καταπολέμηση της φτώχειας όχι όμως για την ε, ενδυνάμωση αλλά για την υποστήριξη για την καταπολέμηση της πείνας και της φτώχειας. Πρέπει όλα τα προσκόμματα και τα εμπόδια να αρθούν, να αντιμετωπιστούν όσον αφορά την κινητικότητα όμως και την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού. Πρέπει από πλευράς του Ευρωπαϊκού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που κάνουμε αυτή τη δουλειά να συνεισφέρουμε. Αλλά με βραδείς ρυθμούς ε, καταφέρνουμε να πετύχουμε να ενδιαφερθούν και να κινητοποιηθούν περισσότερο οι Ευρωπαίοι. Ένα μικρό ποσοστό είναι εκείνο το οποίο εκμεταλλεύεται σήμερα αυτή τη δυνατότητα. Πρέπει να βελτιώσουμε τις δυνατότητες ώστε να τύχουν ε, αυτών των δυνατοτήτων περισσότεροι Ευρωπαίοι. Πώς θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι επαρκή ώστε οι νέοι αλλά και οι ενήλικες να μπορούν να αναλάβουν τον κίνδυνο ως πρωτοβουλία να δημιουργήσουν μια εταιρεία, μια επιχείρηση για να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Από πλευράς των εθνικών πολιτικών πολιτικών ή των ευρωπαϊκών πολιτικών δεν έχουμε τα μέσα που απαιτούνται σε επαρκή βαθμό για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να μπορούν να υποστηριχθούν εκείνοι που θέλουν να ε, ιδρύσουν μια ε, νέα επιχείρηση. Να λάβουμε υπόψη ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσει είναι εκείνε που δημιουργούν τι περισσότερε θέσει απασχόλησης. Κάνουμε λόγο για τι οικογένειε. Πρέπει να ακούσουμε όμω, να εισακούσουμε, να φουγκραστούμε τι λένε οι οικογένειε και ποιε είναι οι απόψει. του. Πολλές προτείνουμε το μέσο χ, ω, το ένα εργαλείο εργαλείο ή το άλλο, όμως πρέπει να ακούμε και να φουγκραζόμαστε τι προσδοκούν οι οικογένειες και ποιες ανάγκες έχουν, πραγματικές ανάγκες σε αυτό τον σημερινό κόσμο. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να μην χτίζουμε κάτι σε ένα διαλυμένο σπίτι και να κάνουμε μερεμέτια. Πρέπει να κάνουμε μια συνολική σφαιρική δουλειά, να ανακαινήσουμε, να αναδομήσουμε, να χτίσουμε εκ βάθρων κάτι καινούριο εκ νέου που θα είναι πραγματικά σημαντικό έργο. Τώρα με το six-pack, την έγκριση των ε, μέτρων για την προώθηση αυτής της πολιτικής, για την ενδυνάμωση της οικονομίας και της πολιτικής μας, ε, είναι σημαντική υπόθεση. Ευχαριστώ, πολύ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Γουαζεύσκη από το Πολωνικό ΣΕΙΜ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είχαμε δύο πολύ, θα έλεγα, χρήσιμες ε, ημέρες συζητήσεων, οι οποίες έδειξαν ότι η δημογραφική κατάσταση και ε, τα κοινωνικά προβλήματα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ποικίλουν από χώρα σε χώρα. Και μάλιστα οι διαφορές μπορεί να είναι και πάρα πολύ μεγάλες. Υπάρχουν χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ο μέσος όρος των εργαζομένων καθορίζεται από νέους μετανάστες οι οποίοι δεν έχουν επαγγελματική εμπειρία και υπάρχουν άλλες χώρες όπως η Εσθονία όπου το τοπίο καθορίζεται θα έλεγα από τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε τομείς όπως ε, η, η κοινωνική πρόνοια, η οποία δημιουργεί, δεν λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ε, που θα ικανοποιούσε τις ανάγκες των εργαζομένων και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων εργαζομένων. Βέβαια, χώρες όπως η Εστονία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν και κάποια κοινά χαρακτηριστικά, γιατί και οι δύο, σαν παράδειγμα, έχουν ε, έλλειψη θέσεων εργασίας και για τους νέους και για τους ηλικιωμένους. Νομίζω λοιπόν ότι το βασικό πρόβλημα είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι θέσεις αυτές αφού δημιουργηθούν θα αποφασίσουμε αν θα πάνε σε ηλικιωμένους ή σε ε, νεότερους ε, υποψηφίους εργαζομένους. Τα πράγματα είναι αλήθεια ότι έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια Υπάρχουν γενικά μεγαλύτερα προσδόκιμα ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ηλικιωμένοι είναι και πιο υγιείς από ό,τι στο παρελθόν, εργάζονται περισσότερο πολλές φορές και παίρνω και τον εαυτό μου σαν παράδειγμα, λέω ο μιλητής. Προσπαθούμε να παραμείνουμε δραστήριοι στην αγορά εργασίας και αυτό είναι ευεργετικό και για, την, και για τα δημοσιονομικά, αλλά και για τους ίδιους ε, τους ε, ηλικιωμένους. Γι' αυτό λοιπόν ε, κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε ας μην προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα μέσο όρο με τα στοιχεία τα οποία έχουμε από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας φτιάξουμε μια εργαλειοθήκη η οποία να περιλαμβάνει πολλές πιθανότητες, δυνατότητες και στοιχεία. Ας μην μιλήσουμε για μια ενιαία στρατηγική, αλλά για ένα σύνολο προτάσεων εύκολα χρησιμοποιήσιμων και στην Εστονία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Ερμάντε Κρό από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του Βελγίου. Α, ε, υπάρχει μια μικρή αλλαγή. θα δώσω πρώτα τον λόγο στον Τζέισον ε, Μουγκλίετ από το Κοινοβούλιο της Μάλτας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αν και η Μάλτα δεν έχει υψηλή ανεργία, έχουμε το πρόβλημα της συμμετοχής στην αγορά εργασίας των γυναικών, των νέων, Ιδιαίτερα για τις γυναίκες άνω των 40 έχουμε πολλά προβλήματα. Έχουν προταθεί αρκετές ε, λύσεις ε, όπως η αύξηση της φροντίδας των παιδιών και εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες ε, και που δίδουν τα κοινωνικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα μου για να προχωρήσει στην κάλυψη των αναγκών αυτών. Το θέμα είναι βέβαια πώς θα αυξήσουμε τις δυνατότητες απασχολησιμότητας, πώς θα δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, πώς δεν θα αποθαρρύνουμε την πρόσληψη εργαζομένων, πώς θα δημιουργήσουμε νέους τύπους εργασίας. Δεν νομίζω, όπως είπε ο κύριος Αγκουστίνο, ότι η λύση στην παγκοσμιοποίηση είναι μια τοπική. Δεν νομίζω ότι μπορούμε μεμονωμένα να καταπολεμήσουμε τις αρνητικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης. Θα πρέπει μοχλεύοντας τις ευρωπαϊκές ικανότητες να καλύψουμε τις ανάγκες που δημιουργούνται στα πλαίσια της απασχόλησης, της απασχολησιμότητας, της παραμονής στην θέση εργασίας και της ενίσχυσης του επαγγελματικού του μέλλοντος και σταδιοδρομίας. Ας βρούμε και τρόπους μείωσης του κόστους παραγωγής, σαν παράδειγμα, της αύξησης της παραγωγικότητας. Στη Μάλτα αυτό είναι ένα θέμα και εδώ οι πολιτικές συνοχής μπορούν να βοηθήσουν. Πώς θα μειώσουμε το κόστος της ενέργειας, σαν παράδειγμα σε χώρες όπως η δική μου, η οποία εξαρτάται κατά 99% από ορυκτά καύσιμα τι κίνητρα μπορούμε να δώσουμε για να καταστήσουμε χώρες όπως τη δική μου ενεργειακά αποδοτικές. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έτσι ώστε να εκμεταλλευτούν πιθανές μειώσεις του κόστους της ενέργειας. Χθες ο κύριος Βανίστελ Ρόι αναφέρθηκε στα θέματα της έρευνας και στα κονδύλια τα οποία δίδονται στην έρευνα και πώς χώρες σύγκλησης και περιοχές σύγκλησης πρέπει να βοηθηθούν έτσι ώστε να επωφεληθούν από την αυξημένη χρηματοδότηση και για την έρευνα. Έτσι ώστε να κερδίσουμε αυτό που ονόμασε ο κύριος Βανίστελ Ρόι ο δρόμος προς την αριστεία. Ε, απαιτείται δυνατότητα, απαιτείται σχεδιασμός και το θέμα δεν είναι μόνο να δούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες της, που ανήκουν στην κατηγορία της σύγκληση, αλλά και ε, περιοχές και χώρες που είναι σε μεταβατική φάση, που σε αυτή τη φάση δεν έχουν όλες τις δυνατότητες παραδοσιακά, δεν έχουν μια μεγάλη παράδοση έρευνας, δεν έχουν μια μεγάλη παράδοση χρηματοδότησης της έρευνας και έχουν και κάποια μειονεκτήματα λόγω του περιφερειακού τους χαρακτήρα, λόγω της γεωγραφικής τους τοποθέτησης. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τις περιφέρειες αυτές έτσι ώστε ε, τα ευρωπαϊκά χρήματα, οι ευρωπαϊκές πιστώσεις να στοχεύουν σωστά και να επιλέγουν σωστά τις περιφέρειες που θα μας επιτρέψει ε, να δημιουργήσουμε τελικά θέσεις εργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Καρίμα Βενελίνοβα Κρούμοβα να πάρει το λόγο από την Βουλή της Βουλγαρίας. Σας ευχαριστώ. Εξ ονόματος της Βουλγαρικής Αντιπροσωπείας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για τη διοργάνωση αυτής της κοινή κοινοβουλευτικής συνάντησης, συνεδρίασης που έχουμε. Η όλο και αυξανόμενη ανεργία, ο πληθυσμός που γυράσκει και είναι υπερήλικος και η ανάγκη των προσαρμογών των κοινωνικών ε, συστημάτων είναι οι προδιαγραφές και οι ε, στόχοι και για τη Βουλγαρία. Πρέπει να τονίσουμε ότι όλα τα προβλήματα παρουσιάστηκαν επειδή υπήρχαν, υπήρξαν χρόνια ολόκληρα αμέλειας και αδιαφορίας. Πρέπει να σχεδιάσουμε για το μέλλον και το μέλλον αυτό να είναι πιο θετικό για μας και τα παιδιά μας. Αναμφίβολα ένα από τα μέσα προς αυτή την κατεύθυνση είναι να αυξηθεί το όριο συνταξιοδότησης ηλικιακά. Χρειαζόμαστε καλύτερα μέτρα ώστε να βελτιωθούν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης. Ξέρουμε ότι δεν θα είναι ταχεία και απλή αυτή η διαδικασία. Γι' αυτό θα θέλαμε να απευθύνουμε έκκληση σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμεριστούν και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές μαζί μας. Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών πάντα βοηθά. Θα πρέπει επίσης να κάνουμε κάπως λόγο και για την αλληλεγγύη. Όσον αφορά την Βουλγαρία θα ήθελα να τονίσω ότι οι Βούλγαροι θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι δεν είναι μόνοι τους και δεν τους έχουν εγκαταλείψει οι άλλοι Ευρωπαίοι. Όσοι είναι πάνω από 60 ηλικιακά θα πρέπει να μπορούν να παραμείνουν στην αγορά εργασίας. Να σας αναφέρω ότι αυτή την εβδομάδα στην, στην Βουλγαρία εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό του 2012. Δεδομένης αυτής της κατάστασης έκδηλης κρίσης, ο προϋπολογισμός μας δημοσιονομικά είναι επαρκής και λαμβάνει υπόψη και τα θέματα τα οποία συζητούμε εδώ, κοινωνική ισότητα και όλα τα άλλα θέματα ως παραμέτρους. Και τα μέτρα τα οποία εγκρίνονται στο ευρωπαϊκό επίπεδο, όλα αυτά θα έπρεπε να υποστηρίζονται και να ε, προωθούνται από όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να εκφράσω αυτές τις απόψεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και τώρα θα λάβει τον λόγο η κυρία Γκούρμαϊ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπω ότι κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας έχουμε αυτή την πολύ σημαντική συνάντηση. Σαν Μιας και προέρχομαι από την Ουγγαρία, θα ήθελα να εκφράσω την χαρά μου που οι Πολωνοί συνάδελφοι οργάνωσαν με τόσο καλό τρόπο τα της Προεδρίας τους. Βλέπω ότι η συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα και θα ήθελα ε, να υπήρχαν πιο συχνές διακοινοβουλευτικές συναντήσεις για τις αλλαγές στην Ευρώπη. Δεν υπάρχουν μόνο οι δημογραφικές αλλαγές, υπάρχει το συνταξιοδοτικό, υπάρχουν τα θέματα της νεότητας, Υπάρχουν ε, πολλά προβλήματα τα οποία γνωρίζει καλά ο Επίτροπος Σάντερ. Έχουμε πολλά εκατομμύρια ανέργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δείτε ότι οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες, θα καταλάβετε ότι έχει σημασία αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μπαρόζο για την ανεργία των νέων ε, και των νέων γυναικών. Γιατί το λέω αυτό. Τον προηγούμενο χρόνο ζήσαμε το λεγόμενο, την λεγόμενη Αραβική Άνοιξη. Μετά πήγαμε στο Τόγκο μετά και, και είδαμε ότι η ανεργία των νέων δεν είναι ένα φαινόμενο αμυγός ευρωπαϊκό, αλλά παγκόσμιο. Και βλέπουμε ότι στην Αφρική η ανεργία των νέων είναι ένα τεράστιο θέμα, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που απειλεί την ειρήνη στην Ήπειρο αυτή. Σχετικά τώρα με, την, με τις μεταρρυθμίσεις του συνταξιοδοτικού, είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σε κάποιες μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό και εγώ είμαι ενοχλημένη από την καθυστέρηση στην κυκλοφορία της Λευκής Βίβλου από πλευράς ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ήταν να κυκλοφορήσει αρχές Νοεμβρίου κανονικά. Πρέπει λοιπόν κάτι να κάνουμε και για το συνταξιοδοτικό σύντομα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτά που θα κάνουμε ε, και την ε, φιλετική διάσταση, γιατί οι γυναίκες είναι πολύ πιο φτωχές από τους άνδρες. Μπορούμε να βοηθήσουμε. Η κυρία Ρέντινγκ, η οποία είναι υπεύθυνη για τα θέματα του φύλου, θα πρέπει να διασφαλίσει την οριζοντιότητα των μέτρων τα οποία θα εφαρμοστούν ε, στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του συστήματος ε, συνταξιοδότησης γιατί αφορά το 50% του κόσμου. Λοιπόν, για τις δημογραφικές αλλαγές θα πρέπει να μιλήσουμε για την προσπάθεια συμφιλίωσης της οικογενειακής ζωής με την επαγγελματική δραστηριότητα. Άκουσα χθε ε, πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες στο συνέδριο του S5 στο Βερολίνο ε, θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να δούμε τι εμπειρίες παίρνουμε από διάφορες χώρες επιτυχημένες και εκτός ίσως Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν χώρες όπου οι γυναίκες είναι ε, σε υψηλό επίπεδο στην αγορά εργασίας με δύο και τρία παιδιά. Η Νορβηγία σαν παράδειγμα είναι ένα καλό τέτοιο παράδειγμα ε, ε, γιατί καλύπτει τις ανάγκες και των παιδιών και των γυναικών και μπορεί κανείς να ζήσει με ικανοποιητικό τρόπο. Έφερα το παράδειγμα της Νορβηγίας, γιατί βλέπουμε ότι και στην Ευρώπη αλλάζουν τα θέματα. Όχι μόνο υπάρχει μια κρίση οικονομική, μια κρίση χρηματοπιστωτική, αλλά και μια θα έλεγα κρίση ηθική και αναφέρομαι στον τρόπο με τον οποίο βλέπει ο λαός την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ ήμουν εισηγήτρια μαζί με τον Αλάλα Μασούρ για την πρωτοβουλία των πολιτών. Πρέπει να εμπλακεί ακόμα περισσότερο ο Ευρωπαίος πολίτης στην προσπάθεια οικοδόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα είναι αν αντιμετωπίζουμε τους πολίτες μας με τον σωστό τρόπο. Έχουμε σωστές επαφές με τους συμπολίτες μας γιατί οι Ευρωπαίοι πολίτες θα ήθελαν να έχουν τη σωστή απάντηση. Λοιπόν, τι θα γίνει να ξέρει ο πολίτης πού θα πάνε τα πράγματα. Ε, οι πολιτικοί πολλές φορές ε, δεν τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει όμως να αγοράσουν παπούτσια για τα παιδιά τους και να διασφαλίσουν το αύριο των παιδιών τους. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ρεαλιστές και πρέπει να είμαστε πραγματιστές. Και γι' αυτό είμαι πεπισμένος ότι όταν συζητάμε τα θέματα αυτά πρέπει να δείξουμε υψηλά επίπεδα ευθύνης. Στην παρούσα φάση όλοι είμαστε ανήσυχοι και όλοι φοβόμαστε τις ευθύνες. Πρέπει να δράσουμε όμως με ταχύτητα και να καταλάβει ο Ευρωπαίος πολίτης ποια είναι η αντίδρασή μας και να καταλάβει ότι είμαστε σε επίπεδο να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκούρμαϊ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο Η κυρία Σκόβα θα λάβει τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα και συγκεκριμένα θα ήθελα να αναφερθώ στην έρευνα και την επιστήμη και την υποστήριξη της ανάπτυξης μέσω αυτών των δραστηριοτήτων. Πρώτα απ' όλα, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την Πολωνική Προεδρία για την επιλογή αυτού του θέματος και την διεξαγωγή αυτού του συνεδρίου. Η κοινωνική συνοχή, το ευρωπαϊκό πρότυπο για την περαιτέρω εξέλιξη ευρωπαϊκά αλλά και παγκόσμια είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Και θα μετρηθεί και πόσο τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να κάνουν κάτι περισσότερο και να μην το αμελήσουν. Ήμουν σε κάθε συνεδρίαση σχεδόν ε, στο κοινοβουλευτικό επίπεδο που παρακολούθησα και λυπούμε για το ότι σήμερα δεν είναι τόσοι παρόντες. Είναι, το θεωρούν ίσως ένα γενικότερο πρόβλημα της ε, Ευρώπης ε, εμείς ε, στην Τσεχία έχουμε πολλές επιφυλάξεις εναντί της ε, Ευρώπης. Αντιμετωπίζουμε αυτές τις επιφυλάξεις και τους δισταγμούς σχεδόν καθημερινά. Οι πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης όταν αναφέρουν την Ευρώπη αναφέρονται σχεδόν πάντα στα κονδύλια των διαθροτικών ταμείων και τις γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις και δυσκολίες. Δεν έχουν το αίσθημα ότι η Ευρώπη μπορεί να τους βοηθήσει άμεσα. Οι περισσότεροι άνθρωποι συμφωνούν όμως όταν λέμε ότι ως σύνολο μόνο η Ευρώπη μπορεί να υπάρξει σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο μπορεί να επιβιώσει μόνο σε ένα ενιαίο ενωμένο σύνολο. Πρέπει να υπερασπιστούμε την Ήπειρό μας, την Ήπειρο της Ευρώπης, την Ήπειρο στην οποία έχουμε το υψηλότερο βιωτικό επίπεδο από πλευράς ευημερίας μια ήπειρο στην οποία προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ευημερία και την αηφορία και πρέπει αυτό να τεθεί μπροστά στην κοινωνική συνοχή και ολοκλήρωση. Είναι ένα όραμα που πρέπει με αυτό οι Ευρωπαίοι να, μπορέσει, να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν τα προβλήματα και να κινητοποιηθούν. Και η κοινωνική συνοχή είναι ένα θέμα που πρέπει ευρωπαϊκά να αντιμετωπιστεί, συνολικά ευρωπαϊκά. Είναι ένα θέμα που αφορά τα κράτη-μέλη, αλλά τα κράτη-μέλη δεν το έχουν έχουν αντιληφθεί ακόμα αυτό όπως πρέπει, ότι είναι ευρωπαϊκό ζήτημα. Θέλω να προσθέσω την φωνή μου στις παρατηρήσεις των άλλων αγοριτών. Τα κονδύλια για την έρευνα και την ανάπτυξη και τις επιστήμες πρέπει να διασφαλιστούν και πρέπει να διοχετεύονται τα κονδύλια όπως γίνεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Αυτό είναι σημαντικό και είναι αρχή που ισχύει για την ε, κοινωνική και ε, συνοχή. Όμως στην ε, Τσεχία τα επιστημονικά ιδρύματα βρίσκονται συνήθως ε, τα περισσότερα σε μία πόλη, σε ένα κέντρο, στην Πράγα και η Πράγα ανήκει στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Τέτοιες περιοχές όπως η Πράγα δεν μπορούν να ζητήσουν να πάρουν κονδύλια από την πολιτική συνοχή και αυτό είναι κρίμα. Θα έπρεπε οι επιστήμονες ε, να υποστηριχθούν ακόμα περισσότερο. Αυτοί βρίσκονται στην Πράγα και πρέπει να υποστηριχθούν. Θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε ένα βέλτιστο επίπεδο και η ανταγωνιστικότητά μας θα μπορούσε να τονωθεί και να ενισχυθεί και θα μπορούσε και η ανάπτυξή μας να προαχθεί, να προωθηθεί όπως πρέπει. Αυτό είναι μια παρατήρηση ε, στο χθεσινό λόγο που εξεφώνησε ο κύριος Φανίστελ Ρόι. Ένα παρόμοιο πρόβλημα πιστεύω ότι αντιμετωπίζουν και άλλα μικρότερα κράτη-μέλη όπως και εμείς οι Τσέχοι. Και μια επιθυμία που θα ήθελα να εκφράσω για το 2012. Εύχομαι στο Εθνικό Κοινοβούλιο και στα, ε, στα Εθνικά Κοινοβούλια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ορίσουμε ένα νέο όραμα. Νέο όραμα για μια νέα Ευρώπη. Και έτσι να συνεισφέρουμε από πλευρά μα για μια ειρηνική ανάπτυξη και ευημερία και αηφορία για το μέλλον. Για το μέλλον τη Ευρώπη. Και ελπίζω και πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε από κοινού. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Χόπκινς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, πράγματι η παρουσίαση την οποία έκανε και η κυρία Γκορμάη από την Ουγγαρία είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον λόγω της, ε, του θέματος ε, της ανεργίας που έφυξε και των κοινωνικών προβλημάτων που δημιουργούνται από την ανεργία. Κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανησυχούν για χαμηλά ποσοστά γεννητικότητας. Εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν το έχουμε αυτό. Έχουμε ίσως ε, υψηλά επίπεδα γεννητικότητας και έχουμε και υψηλά ποσοστά μετανάστευσης. Ακόμα και από τις χώρες με χαμηλή γεννητικότητα βλέπουμε οι νέοι να φεύγουν και να πηγαίνουν σε άλλες χώρες όπως η Βρετανία. Αυτό είναι κάτι το οποίο ίσως εκπλήσει. Εμείς θέλουμε φυσικά τους εργαζομένους με ικανότητες να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της δικής μας χώρας, αλλά αφήνουν τη δική τους χώρα, δημιουργούνται προβλήματα, δημιουργούνται κενά και στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε πάρα πολλά προβλήματα με τους ηθαγενείς εισαγωγικά νέους οι οποίοι παραμένουν άεργοι ε, διότι κοστίζουν περισσότερο. Λοιπόν, οι θέσει εργασίας τις οποίες θα μπορούσαν να καλύψουν πηγαίνουν στις πολύ εντυπωσιακές στους πολύ εντυπωσιακούς τίτλους και περγαμηνές των εργαζομένων που προέρχονται από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πράγματι αν όλα τα προσόντα των εργαζομένων που έρχονται στη χώρα μας από άλλες χώρες είναι τόσο εντυπωσιακά, πράγματι οι χώρες σας είναι πάρα πολύ τυχερές. Ε, ομιλούν εξαιρετικά την αγγλική γλώσσα σαν παράδειγμα, ενώ εμείς οι Άγγλοι δύσκολα μιλάμε, έστω και ψήγματα άλλης γλώσσας. Εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα της ανεργίας είναι σαφές και οι μεγάλες μετακινήσεις των πληθυσμών δεν θα λύσουν το πρόβλημα της ανεργίας όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά στον κόσμο γενικότερα. Επίσης τα προβλήματα τα οικονομικά δεν θα επιληθούν από ε, μέτρα λιτότητας. Τα μέτρα λιτότητας ε, δημιουργούν υψηλότερη ανεργία, χαμηλότερα έσοδα, αυξημένο κοινωνικό κόστος και χειροτερεύουν την κατάσταση. Δεν είναι σωστός ο τρόπος των περικοπών για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα λοιπόν. Είναι σαφές ότι θα πρέπει στις χώρες μας να ζούμε ανάλογα με τα μέσα που έχουμε και τις δυνατότητές μας, αλλά να εκμεταλλευόμαστε ταυτόχρονα και όλες τις ευκαιρίες και δυνατότητες τις οποίες έχουμε. Αν συνδυάσουμε την παραγωγικότητα με την ικανότητα του εργατικού δυναμικού, τότε θα μειώσουμε την ανεργία, θα βελτιώσουμε τα επίπεδα ζωής και θα μειώσουμε και ε, το ε, δημοσιονομικό έλλειμμα. Τώρα δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά υπάρχει μια ολόκληρη σειρά μέτρων τα οποία θα πρέπει να πάρουμε. Νομίζω ότι ο αποπληθωρισμός ο οποίος απασχολεί τόσο πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες προχωρημένες χώρες, είναι βασικός στόχος, ενώ θα πρέπει να αναπληθωρήσουμε. Ξέρουμε τι έγινε στις αρχές του 30, όπου οι χώρες έκοψαν τις θέσεις απασχόλησης, δημιουργήθηκαν ε, τεράστια ποσοστά ανεργίας και μόνο μέσω των κεινσιανών πολιτικών στα τέλη της δεκαετίας του 30 τα πράγματα κάπως βελτιώθηκαν. Ας μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος λοιπόν. Ας διασφαλίσουμε ένα λογικό πρότυπο κοινωνικής συνοχής. Ας αλλάξουμε σωστά τη διαχείριση της οικονομίας προς το συμφέρον των πολιτών και να μην εγκαταλείψουμε τα πάντα στις διαθέσεις των αγορών που δεν λύνουν τα προβλήματα. Είναι της μόδας οι αγορές. Αλλά βλέπουμε ποια είναι τα προβλήματα των οικονομιών των αγορών. Βλέπουμε ότι καλό θα ήταν να μπορούσαμε να δημιουργήσουμε την πλήρη απασχόληση. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Θα πρέπει να είμαστε παρεμβατικοί και να μην αφήσουμε την αγορά ανεξέλεγκτα να ρυθμίζει τα πάντα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η Έντις Μπάουερ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εισαγωγικά θα ήθελα να εκφράσω όλη μου την ευγνωμοσύνη στην Πολωνική Προεδρία που έθεσε στην ημερήσια διάταξη αυτές τις κοινωνικές θεματικές διότι έχω την εντύπωση ότι φέτος σε αυτό το σώμα δεν συζητήσαμε καθόλου για κοινωνικά θέματα. διότι δηλαδή, ό,τι δεν συζητήσαμε σε ένα χρόνο, το συζητήσαμε δύο μέρες σε αυτή τη συνάντηση. Ξέρουμε ότι την πρωτοκαθεδρία στις συζητήσεις μας την είχαν η οικονομική και κοινωνική κρίση. Έφτασε όμως η στιγμή να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένα κοινωνικό πρόσταγμα, ένα κοινωνικό κατεπήγον, μια κρίση αξιών, το οποίο είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένο με την οικονομική και κοινωνική κρίση. Ως προς την ανάλυση Έχουμε εμεί στη διάθεσή μας μέσα, ε, επαρκέστατα μέσα, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά το να το κάνουμε είναι το δύσκολο. Και πάντα περισσότερο συνειδητοποιούμε και βλέπουμε ότι αυτό συμβαίνει και για τα περισσότερα προβλήματα που είναι τόσο διαφορετικά. Όσον αφορά τώρα τη δημογραφική κρίση, εκκινώντα από αυτή την αρχή και αυτή την αφετηρία, να δώσω ένα παράδειγμα. Εμεί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχουμε τόσε πολλέ δυνατότητε στη διάθεσή μα για την αύξηση φυσικά του ποσοστού γεννήσεων της γεννητικότητας. Ένα μέσο υπάρχει. Είναι η γονεϊκή άδεια των μητέρων, η, νομοθεσία υπέρ της μητρικής άδειας. Οι ειδήσει όμως τα μαντάτα από το Συμβούλιο δείχνουν ότι αυτή η πρόταση που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το Συμβούλιο δεν γίνεται, δεν γίνεται δεκτή. Και αυτή η πρόταση θα αντιμετωπιστεί με αρνητικό τρόπο. Θα είναι μια ήττα αυτό τι δείχνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο βλέπετε να υιοθετηθούν έστω και ελάχιστες προδιαγραφές για τις λύσεις εκείνες που έχουν σκεφτεί ήδη τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν και να μην ξεχνάμε ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στον κοινωνικό τομέα δεν έχουν αρμοδιότητες να νομοθετήσουν καθοριστικά. Έχω τον λόγο και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω την κιανή κάρτα, την μπλε κάρτα και δράτω με τις ευκαιρίες να σας ρωτήσω πώς έχει η σημερινή κατάσταση, τι γίνεται με την νομοθετική πρόταση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο όσον αφορά την μητρική άδεια, γονεϊκή άδεια. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το μπαλάκι θα περάσει στην πλευρά του, στο γήπεδο του Ευρωκοινοβουλίου ή τι θα γίνει. Όσον αφορά την ενεργογύρανση έχουμε πάλι ένα πρόβλημα εδώ ενώπιον μας που ίσως δεν είναι σημερινό πρόβλημα αλλά είναι αυριανό πρόβλημα σίγουρα και μια και είναι το πρόβλημα του μέλλοντος, αυριανό πρόβλημα, θα πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις ε, στο διάστημα που έχουμε τώρα στη διάθεσή μας. Αναφέρατε πρόεδρε προηγούμενα ότι ένα συγκεκριμένο ποσοστό ενεργοποιείται μόνο μόνο. Αν δούμε το ποσοστό των γυναικών 37% είναι αυτό το ποσοστό και αυτό δείχνει ότι δεν γυράσκουμε με τον ίδιο τρόπο. Οι γυναίκες γυράσκουν νωρίτερα και με άλλες ε, ταχύτερες ε, διεργασίες. Ε, βρίσκονται σε διαφορετική θέση λοιπόν και πάλι σε σχέση με τους άντρες. Λοιπόν πάλι μέσα σε αυτό το πλαίσιο αξίζει για άλλη μία φορά διπλάσια να αφιερώσουμε τις προσοχές μας σε αυτό το θέμα, την προσοχή μας σε αυτό το θέμα. Το μεδούλι, την ίδια την ουσία του θέματος. Όταν πρόκειται για περίοδο κρίσης και έχουμε θέματα γυναικών και δικαιωμάτων και ισότητας των γυναικών πρέπει σε βάθος να τα δούμε σε όλες τις παραμέτρους διότι έχουν πολύ ε, σημαντικές επιπτώσεις στην εμβέλειά τους. Και ένα δεύτερο θέμα όσον αφορά την μείωση του ποσοστού φτώχειας, την αντιμετώπιση της φτώχειας από πλευρά μας. Όλοι γνωρίζουμε ότι από τότε που εγκρίθηκε η στρατηγική για το 2020 συμφωνήσαμε όλοι και για την μείωση του ποσοστού φτώχεια. και της φτώχειας γενικά και βλέπουμε ότι το αντίθετο συμβαίνει. Οι φτωχοί στην Ευρώπη αυξήθηκαν 20 εκατομμύρια παιδιά ζουν σε καθεστώς φτώχεια στην Ευρώπη σήμερα. Διατίθεται το ερώτημα τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι και αυτό έχει ευρύτατες ε, κοινωνικές επιπτώσεις στην εμβέλειά τους, διότι το μελλοντικό ανθρώπινο δυναμικό με αυτόν τον τρόπο μειώνεται, συρρυκνώνεται. Είναι το ανθρώπινο δυναμικό που πρέπει και θα έχει η Ευρώπη στο μέλλον. Δεν μπορούν αυτά τα παιδιά να μορφωθούν και να καταρτιστούν. Μιλήσατε και κάνατε λόγο για το ότι οι διαφορές ε, επιδεινώνονται και αυξάνονται. Και αυτό συμβαίνει πράγματι. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Η κοινωνική ψαλίδα ανοίγει όλο και περισσότερο και οι διαφορές εντείνονται όλο και περισσότερο. Ένας ιστορικός είπε κάποτε ότι οι διαφορές όσον αφορά τους μισθούς και τα κοινωνικά θέματα ήταν πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με την περίοδο της, ε, πριν από τον ε, πόλεμο και μετά τον πόλεμο. Πώς μπορούμε να λύσουμε αυτές τις μεγάλες διαφορές. Ξέρουμε ότι υπάρχουν τεράστιες κοινωνικές εντάσεις ε, που μπορούν να δημιουργούνται από αυτές τις κοινωνικές ανισότητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Στην εκπρόσωπο της Εσθονικής Βουλής έχετε το λόγο. Eh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Τα πράγματα εξελίσσονται άσχημα. Ομολογώ ότι είμαι ε, ανήσυχη. Ίσως ε, χτες και σήμερα σε ό,τι είπα φάνηκα λίγο υπερβολική. Ίσως να έδωσα και την εντύπωση ότι η Εσθονία δεν έχει πετύχει και πάρα πολλά πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πάμε άσχημα. Ο κύριος Μπούζαγκ είχε έρθει στη Βουλή της Εστονίας πρόσφατα και μας συνεχάρει για τις προσπάθειες τις οποίες κάνουμε. Το θέμα είναι πώς βλέπει κανείς τα πράγματα. Εγώ είμαι αρκετά αισιόδοξη. Νομίζω ότι έχουμε πετύχει αρκετά στον τομέα τον κοινωνικό και για τα υπόλοιπα θέματα τα οποία απασχολούν τους εστονούς. Σαν παράδειγμα η γονική άδεια οι γυναίκες παίρνουν σαν παράδειγμα μέχρι και 16 μήνες έμιστης άδειας. Γενικά υπάρχουν βελτιώσεις στην κοινωνική κάλυψη. Έχουμε το αντίστοιχο πρόγραμμα με την Πολωνία 60 συν, 60 και. Προσπαθούμε να μην αποκλείσουμε από την αγορά εργασίας τους ηλικιωμένους και πολλές φορές κάποιοι δεν καταφέρνουν καν να επωφεληθούν από τις συντάξει τους γιατί δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια. Πηγαίνουν όπως λέμε από τη δουλειά στον τάφο. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά και εξαρτώνται εν πολλής ε, από τη δημοσιονομική πολιτική. Η δημοσιονομική πολιτική μας ήταν η καλύτερη μας είχαν πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά Τύχει όμως και υψηλό τίμημα και το τίμημα το πληρώσαμε. Η ζωή, η καθημερινότητα είναι δύσκολη και αυστηρή. Η μεγαλύτερη οικογένεια που έχουμε στην Εστονία με 16 παιδιά πραγματικά πολύτεχνοι μετανάστευσαν στο Ηνωμένο Βασίλειο γιατί ζουνε καλύτερα εκεί με τόσα παιδιά. Είναι περίεργο αυτό, όπως είπα ήταν η μεγαλύτερη οικογένεια πολυτέκνων την οποία είχαμε και τη χάσαμε. Ε, ξεκινήσαμε συγκεκριμένα προγράμματα για την υποστήριξη των ιατρών, οι οποίοι ε, πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες ε, των περιοχών οι οποίες εγκαταλείπονται από τους κατοίκους τους. Τους πληρώνουμε 15.000 ευρώ το χρόνο ε, σε, για να καλύψουν τις ανάγκες αυτές. Βέβαια στη Φιλανδία 15.000 ένας γιατρός θα πάρει σε 2-3 μήνες και γι' αυτό οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε είναι γνωστές. Είναι δυσκολίες οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και μέσω της πολιτικής συνοχής και θα πρέπει ε, τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά να διανέμονται με τον σωστό τρόπο. Ποτέ δεν θα είναι όλοι ικανοποιημένοι βέβαια. Οι νέες χώρες έχουν προβλήματα χρηματοδότησης, οι παλαιές χώρες έχουν προβλήματα υπογεννητικότητας. Αύριο θα έχουμε και άλλα προβλήματα ίσως. Εγώ σαν αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της χώρας μου δεν μου αρέσει ο προϋπολογισμός που καλούμεθα να ψηφίσουμε αύριο μεθαύριο, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να βοηθήσουμε και να λύσουμε τα προβλήματα. Πρέπει να βοηθήσουμε και με τη συνεισφορά μας τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Τα πάντα, όλα τα μέτρα έχουν ένα κόστος, έχουν ένα τίμημα και το τίμημα αυτό είναι μερικές φορές δυσβάστακτο, ας είμαστε ειλικρινείς. Ε, ευχαριστώ πολύ για αυτήν την εύστοχη παρατήρηση. ο Λαϊός μίλε από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, αυτές τις τελευταίες δύο ημέρες ε, διαφορετικά θέματα δείξαμε και καλύψαμε δημογραφικές αλλαγές στην Ευρώπη, τα θέματα μετανάστευσης, την κατάσταση των γυναικών στην αγορά εργασίας, την κατάσταση των νέων, την κατάσταση των ηλικιωμένων. Όμως, βρήκαμε έναν παρονομαστή. Κάθε αγορητής ανέφερε και είπε ότι ανησυχεί για το ευρωπαϊκό πρότυπο, για τις αρχές και αξίες της Ευρώπης ως κοινωνικού προτύπου, για το πρότυπο της κοινωνίας ευημερίας που ε, υπονομεύεται ή απειλείται. Κάναμε λόγο για όλα αυτά τα πράγματα. Κάποια στοιχεία θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στα εξής. Όταν κάνουμε λόγο για τις γυναίκες στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να δούμε και να πούμε ότι εφόσον συνεχίζουν και υπάρχουν αντιφάσεις και αντιθέσεις όσον αφορά την επαγγελματική ζωή και την οικογενειακή ζωή για τις γυναίκες θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα που θα, θα αντιμετωπίζουμε. Η συνέπεια αυτής της αντίφασης είναι ότι οι γυναίκες όλο σε μεγαλύτερη ηλικία τεκνοποιούν, γίνονται μητέρες. Αυτό έχει επιπτώσεις και στο δημογραφικό επίπεδο και στο κοινωνικό επίπεδο. Εφόσον αυτές τις αντιθέσεις ε, ή όσον αφορά το πρόβλημα της σύγκλησης, της ε, συμφιλίωσης, του συνδυασμού της επαγγελματικής ζωής με την οικογενειακή ζωή δεν επιλύουμε το πρόβλημα, θα συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε πρόβλημα και συνέπειες του. Αναφέρθηκε και η εκπαίδευση, κατάρτιση μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Ένα παράδειγμα θα ήθελα να αναφέρω και με το παράδειγμα αυτό θα ήθελα να καταδείξω ποια προβλήματα αντιμετωπίζουμε όσον αφορά τους νέους και όσον αφορά και τους ηλικιωμένους. Ξέρουμε ότι στην Ουγγαρία έχουμε το πρόβλημα ότι ο τομέας της εκπαίδευση και της παιδείας και της αγοράς εργασίας αντιμετωπίζουν προβλήματα. Για τους νέους η σταδιοδρομία όσον αφορά την ε, διδασκαλία δεν είναι θελκτική. Θα πρέπει να δημιουργηθεί προοπτική και δυνατότητες για τους νέους. Όμως αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή το πρόβλημα το μισθολογικό. Πώς δηλαδή το μισθολογικό πρόβλημα σε αυτό τον τομέα θα μπορούσε να επιληθεί και να αντιμετωπιστεί. Αν θέλουμε να είναι πιο θελκτική αυτή η σταδιοδρομία πρέπει να προσφέρουμε ικανοποιητικούς μισθούς σε εκείνους τους νέους που θα ακολουθήσουν αυτή την σταδιοδρομία, αυτή την καριέρα. Όμως δημιουργούνται επειδή υπάρχει υποτίμηση του έργου όσον αφορά τους ε, δασκάλους μια και άλλοι κερδίζουν πολλά περισσότερα χρήματα και έχουν πολύ μεγαλύτερους μισθούς με άλλες δραστηριότητες από εκείνους ε, και μάλιστα και σε νεότερη ηλικία. Πρέπει μεγάλες προσπάθειες να γίνουν για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Διαφορετικά θα έχουμε εντάσεις, εντάσεις και τριβές αυτές ακριβώς που θέλουμε να καταπολεμήσουμε. Όλοι ανησυχούμε για το μέλλον του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας ότι όχι μόνο η Ευρώπη βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο αλλά παγκόσμια όλος ο κόσμος συνολικά οικουμένη και πρωτοβουλίες ε, για μια ευρασιατική, ευρωασιατική ένωση όπως κάποιοι προτείνουν να ακολουθηθεί. Πίσω από τέτοιες ε, ε, προτάσεις υποκρύπτονται φυσικά ρωσικές και άλλες φιλοδοξίες. Πρέπει όμως να έχουμε υπόψη μας ότι έχουμε και νέους ανταγωνιστές, νέους εταίρους, νέους τομείς. Σε αυτόν τον τομέα ανταγωνισμού δεν έχουμε μόνο την οικονομική κρίση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αλλά και άλλους εμπλεκόμενους στην αγορά που μας ανταγωνίζονται, άλλους που δεν είχαμε και δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε ακόμα τις επιπτώσεις στο μέλλον από πλευρά τους. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Άντρεϊ Γκρίπ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Σε αυτήν εδώ τη συνάντηση και στην ανταλλαγή απόψεων για κοινωνικά θέματα και δημογραφικά προβλήματα, όπως επίσης και για την αηφορία, όλα αυτά εντάσσονται μέσα σε ένα πλαίσιο. 8 και 9 του μηνός θα έχουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. για το οποίο θα πρέπει να βρούμε και μία λύση για την κατάσταση του ευρώ. Θα πρέπει κατά αυτόν τον τρόπο να ρυθμίσουμε την κατάσταση 17 κρατών μελών στο μέλλον, ούτω ώστε να υπάρχει δημοσιονομική συνοχή χωρίς να υποσκάψουμε το ευρώ. Και υπάρχει και μία, ένας φυσικός πειρασμός, που είναι να κάνουμε οικονομίες. Πού μπορούμε να κάνουμε εμείς οικονομίες? Στις κοινωνικές δαπάνες. Στη συζήτηση που είχαμε σήμερα και όπου συζητήσαμε το πόσο σημαντική είναι η κοινωνική συνοχή, είπαμε ότι ναι, χρειάζονται δαπάνες αλλά και ορθολογικότητα. Είπαμε ότι η λύση δεν ε, επαφίεται μόνο στις περικοπές. Το κοινοβούλιο είναι ο κατάλληλος τόπος για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Πολύ συχνά στην εκλογική μου περιφέρεια Σύναντο, κόσμο, παράδειγμα φοιτητέ που μου λένε «Μα πού είναι η κοινωνία σε όλα αυτά» Μόνο για αγορές μιλάμε, για, για, για χρηματοπιστωτικές αγορές. Πού είναι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, η κοινωνία. Βάσει ποιου εμείς αποφασίζουμε τις πολιτικές μας. Πρέπει να ακούσουμε εμείς αυτό το μήνυμα, να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Και να πούμε ότι ναι, δεν ασχολούμαστε μόνο με χρηματοπιστωτικές αγορές, αλλά και με το γεγονός ότι θέλουμε να βελτιώσουμε την ευημερία των Ευρωπαίων. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Διότι κατά την τελευταία συζήτηση που είχαμε, για τον προϋπολογισμό του 2012 καταλήξαμε σε έναν συμβιβασμό όπου τα κράτη-μέλη είπαν ότι δεν θα δώσουν την... <coughs> Δεν θα δώσουν το ποσοστό το οποίο θα έπρεπε να έδιναν στο κοινωνικό ταμείο, αλλά ότι θα, αναδια... θα πρέπει να επαναδιαμορφώσουν την δαπάνη. Εξάλλου, όπως είπε και ο Επίτροπος και ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου, θύμισαν τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Και αυτό το οποίο μου είχε αρέσει εμένα ιδιαίτερα στη στρατηγική 2020 ήταν ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε όπου εγκαταλειπόταν η τεχνοκρατική παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλούσαμε για κοινωνικό αποκλεισμό, για την καταπολέμησή του. Εμείς θα πρέπει να δράσουμε στον τομέα της παιδείας για παράδειγμα γιατί τι κάνουμε εμείς με όλους αυτούς τους νέους που δεν τελειώνουν τις σπουδέ τους, πώς θα βρουν αυτή η δουλειά, πώς θα τους δώσουμε απασχόληση όταν την βασική, δεν τελειώνουν τους, τους κύκλους της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Το 15% των νέων στην Ευρώπη υπάρχουν παράγοντες οικογενειακοί, κοινωνικοί. Ρωτώ λοιπόν, Επίτροπε, Μήπως τελικά αυτό το τόσο μεγαλόπνο σχέδιο της Ευρώπης του, 2020, του 2020 να ξεχαστεί, να μην ασχοληθεί με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, στην ψηφιακή αγορά, στην υγεία, στις κοινωνικές δαπάνες, στην παιδεία. Δεν θα έπρεπε να ξαναδείτε εσείς το δημοσιονομικό πλαίσιο αυτού του σχεδίου, το οποίο έχει ως στόχο το ξεπέρασμα του κοινωνικού αποκλεισμού. Για την ευρωπαϊκή συνεργασία μίλησε ο Επίτροπος Μπαρνιέ ο οποίος θύμισε ότι μέχρι το 2020 αυτές οι επιχειρήσεις θα δημιουργήσουν 5.000 θέσεις εργασίας. Στη βάση αυτών των προοπτικών δεν θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας και όλους αυτούς τους κοινωνικά αποκλεισμένους και να ξεκινήσουμε σχέδια κοινωνικών συνεταιρισμών διότι υπάρχουν εμπειρογνώμονες μεν αλλά μας λείπουν επαΐοντες στα οικονομικά που θα μας επέτρεπαν να λύσουμε σε τοπικό επίπεδο ε, κάποιο πρόβλημα. Ο γερουσιαστής Αουγκοστίν είπε «Μα πόσα λεφτά ξοδεύονται στην Πολωνία για κοινωνικές παροχές». Εγώ φαντάζομαι ότι ανατρέποντας αυτή την τάση, εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είμαστε αυτοί που θα δίνουμε την πετονιά και όχι το ψάρι. Όλοι είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά το κέντρο όλων αυτών είναι η κοινωνία. Ευχαριστώ. Ο εκπρόσωπος της Πορτογαλικής Βουλής έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε πίτροπε αγαπητοί συνάδελφοι, σε σχέση με την παρέμβασή μου, ε, ήθελα προηγούμενα να αναφερθώ σε αυτές τις δύο ημέρες εργασίας που δείχνουν σαφώς ε, ότι οι απόψεις των διαφορετικών κοινοβουλίων είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση όσον αφορά την πολυμορφία και την πολυπλοκότητα της Ευρώπης που σε όλα τα θέματα πρέπει να προσπαθούμε να βρούμε απαντήσεις μέσα από αυτήν στην Ευρώπη. Στην παρέμβαση επί της ουσίας ε, θα ήθελα να αναφερθώ στο εξής. Αυτές τις δύο ημέρες επικεντρωθήκαμε και συζητήσαμε την υποστήριξη που μπορούμε να δώσουμε για την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, στην ε, μητρότητα και τον συνδυασμό της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή. Ε, το πρότυπο το κοινωνικό της Ευρώπης που πρέπει να κερδίσουμε ως στίχημα. Όμως σε αυτές τις πολιτικές η ύπαρξη του κοινωνικού προτύπου χρειάζονται όλες αυτές ε, οι ανάγκες χρηματοδότηση, κονδύλια, μεγάλους πόρους, πολλούς πόρους. Υπάρχει κατεπίγουσα ανάγκη να αποφασιστεί ποιο θα είναι το μέλλον του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου και πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτό για παράδειγμα, από πλευρά ε, τη ε, Επιτροπή, ε, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, στην οποία ανήκω στην Πορτογαλική Βουλή, εξετάζει αυτά τα θέματα και όλο και περισσότερο βλέπουμε ότι η ύπαρξη αυτών των πλαισίων απειλείται. Υπάρχουν σημαντικέ περικοπές στον προπολογισμό τη Πορτογαλίας, ακριβώ στην εκπαίδευση και στην υγεία, που είναι θεμελιώδει πυλώνε για αυτά που συζητούμε εδώ από πλευρά επενδύσεων και κονδυλίων. Υπάρχουν εδώ εδώ αντιφάσεις για θέματα τα οποία συζητούμε εδώ, για την πολιτική συνοχή, για την αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών και την διασφάλιση του κοινωνικού προτύπου της Ευρώπης και μετά των μέτρων που λαμβάνονται καθημερινά από τα κράτη-μέλη και τις κυβερνήσεις τους με περικοπές, περικοπές και όλο και μεγαλύτερη λιτότητα. Είναι αναγκαίο λοιπόν οι ηγέτες της Ευρώπης να κάνουν μια σαφή αναμφίσιμη επιλογή. Θέλουν να διατηρήσουν ή όχι το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο ως αρχή, πολιτισμική αρχή και θεμέλια της ε, ε, πρότασης της Ευρώπης. Με τις ε, αλλαγές αυτές τις δημογραφικές πώς θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τη διασφάλιση αυτού του προτύπου. Πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε και να χρηματοδοτήσουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο. Αυτό είναι το ερώτημα. Εγώ πιστεύω ότι είναι δυνατόν να διατηρηθεί σήμερα και στο μέλλον το ευρωπαϊκό κοινωνικό αυτό πρότυπο. Μόνο που χρειάζεται να γίνουν επιλογές και αναλυθούν αποφάσεις με σαφή αναμφίσιμο τρόπο και γοργά, γρήγορα. Οι πολιτικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν έχουν κατεπήγοντα χαρακτήρα. Γι' αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον Επίτροπο που βρίσκεται εδώ παρόν θα ήθελα να μας καθησυχάσει και να μας πει μερικά λόγια που θα δείχνουν την προοπτική στο μέλλον. Ευχαριστώ. E, Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας και τώρα θα λάβει τον λόγο ο κύριος Επίτροπος, ο κύριος Λάσλο Άντορ, παρακαλώ. Αξιότιμοι βουλευτές κυρίες και κύριοι, πρέπει να ζητήσω συγγνώμη για μια πολύ σύντομη απάντηση που θα δώσω, γιατί κράτησε πολύ περισσότερο αυτή η συνεδρίαση από ό,τι προβλεπόταν και θα έπρεπε τώρα να βρίσκομαι σε μια άλλη διάσκεψη για θέματα ανισότητας. Και όμως με ένα σύντομο τρόπο θα ήθελα να, να διασφαλίσω σε κάποιους από εσάς στην κυρία που υπογράμισε τη σημασία των θεμάτων ανισότητας για παράδειγμα στον, στη σημερινή ευρωπαϊκή κατάσταση και να μην αφήσουμε τα πράγματα απλά στις αγορές και στις οικονομικές πολιτικές για την ε, αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων χωρίς ε, επαρκή προσοχή στην κοινωνική διάσταση και τις κοινωνικές ανάγκες. Με τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, στην οποία νομίζω αναφέρθηκαν και υποστήριξαν τα περισσότερα σχόλια και οι παρατηρήσεις σας, υπάρχει ένας σαφέστατος στόχος και ένα σύνολο πρωτοβουλειών και δράσεων. Όχι μόνο να διατηρηθεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο, αλλά να ενισχυθεί, να ενδυναμωθεί ακόμα με πολιτικές για την απασχόληση και την καταπολέμηση της φτώχειας. Το πρόβλημα είναι ότι ταυτόχρονα υπάρχει και μια κρίση χρέους, υπερχρέωσης, μια χρηματοοικονομική, δημοσιονομική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζήτημα που τίθεται αυτή την εβδομάδα, εβδομάδα λήψεως αποφάσεων αλλά και πέρα από αυτήν για το μέλλον, η χρηματοοικονομική κρίση έχει επιπτώσεις ε, με πολλούς τρόπους ε, και θα έπρεπε να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε ώστε το δυναμικό των χωρών μας να ενδυναμωθεί, να διασφαλιστεί και να διασφαλιστεί και η ε, συνεκτικότητα του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου δεν είναι μόνο το ευρώ το νόμισμα το οποίο κινδυνεύει και διακυβεύεται, είναι η ίδια η κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη και το ίδιο το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο λοιπόν. Αλλά μετά στη συνέχεια θα πρέπει να επιλεγούν σωστά οι πρωτοβουλίες και ε, προτεραιότητες από πλευράς Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Άκουσα τον εκπρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου ότι είναι, λέει, έχει αιμονές ε, η ιδέα πρέπει να δούμε ποιος είναι ε, που έχει αιμονές και είναι αιμονικός όσον αφορά κάποια θέματα όπως ε, θέματα ε, στασιμοπληθωρισμού και άλλα. Βλέπουμε ότι εδώ το θέμα του πληθωρισμού και αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερο πρόβλημα από ίσως τη μεγαλύτερη χώρα, η ισχυρότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έπρεπε να προσαρμοστούν οι προσπάθειές μας να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα χρήματα με το σωστό τρόπο και όχι να έχουμε αιμονές. Είναι σαφές ότι με την πειθαρχία, την λιτότητα, τις κυρώσεις αυτή η κρίση δεν θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Η κρίση μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο αν υπάρχει και διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο αλληλεγγύης και υψηλό επίπεδο συντονισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Και έτσι πρέπει να αναλάβει και να διαδραματίσει ένα ουσιώδη σημαντικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλα αυτά. Οι συζητήσεις κατέδειξαν ότι περισσότερα πρέπει να γίνουν ώστε να επεξεργαστούν εξηγηθούν ε, οι επιπτώσεις αυτού του ε, πολύπλοκου πλαισίου και ο ρόλος των δημοσιονομικών ε, πρωτοβουλειών και δράσεων των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Αυτό ισχύει και για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο επίσης, διότι το γεγονός ότι προτείναμε κατόφλι, συγκεκριμένο κατόφλι για τα μέτρα κοινωνικής ένταξης και ολοκλήρωσης δεν είναι μόνο παθητικά μέτρα, είναι μέτρα ολοκλήρωσης και κοινωνικής ένταξης ενεργά, Συμπεριλαμβάνουν και την ένταξη των ατόμων με ειδικέ ανάγκε ή ε, μειονεξίε, του Ρωμά, του Τσιγκάνου, ε, να μπορέσουν και αυτοί να ενταχθούν στην αγορά εργασία ε, και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματά τους. Η υποστήριξη της εκπαίδευσης, παιδείας, κατάρτισης για τους πιο ευάλωτους και για τους νέους είναι κάτι που πρέπει να το δούμε υπό το πρίσμα της μελλοντική απασχολησιμότητας. Δεν αποσυνδέονται όλα αυτά από την αγορά εργασίας ή από το δυναμικό της ε, ε, ευρωπαϊκής οικονομίας ε, και για το μέλλον. Επιπλέον έχουμε περαιτέρω μέτρα και εργαλεία για να δραστηριοποιηθούμε. Για παράδειγμα, ε, το πρόγραμμα για την, ε, ε, τις μικροεπενδύσεις που λειτουργεί θετικά, αλλά και άλλες πηγές και δυνατότητες όσον αφορά τα ευρωπαϊκά κονδύλια το πρόγραμμα για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας του επιχειρήν γενικότερα που μπορεί να, είναι, να αποβεί ε, θετικό για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης και υπέρ των νέων. Και να αντιμετωπιστεί και η ανεργία των νέων, που η ανεργία των νέων είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά τα κοινωνικά θέματα, τις κοινωνικές υποθέσεις πανευρωπαϊκά. Κυρίες και κύριοι, θα μπορούσα να συνεχίσω αυτή την απαρίθμηση ε, των εμπειριών και βιωμάτων μας, ε, αναφέροντας για παράδειγμα και τα στοιχεία σε σχέση και με το λευκό βιβλίο όπως συζητήθηκαν και αναφέρθηκαν από την κυρία Γκούρμαϊ. Αλλά θα ήθελα να ολοκληρώσω εδώ μετά από αυτές, αυτή την παρέμβασή μου. Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να έχουμε, επικοδομητικές, ε, να έχουμε επικοδομητική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Φυσικά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων για την ενεργή του συμμετοχή στη συζήτηση. Δίνω το λόγο στον Υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων της Πολωνίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους σας για όλα αυτά τα σχόλια που κάνατε στη συζήτηση. Ευχαριστώ. γιατί οργανώσατε υπό Πολωνική Προεδρία αυτήν την διάσκεψη για την κοινωνική πολιτική και τα δημογραφικά προβλήματα. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος όταν ακούω την κυρία Μπάουερ για την οδηγία σχετικά με την μητρότητα. Η Πολωνική Προεδρία προσπάθησε να κάνει ό,τι μπορεί για να συνδυάσει οικογενειακή ζωή με την μητρότητα. Ήμασταν ιδιαίτερα δυναμικοί σε αυτόν τον τομέα. Στην Κρακοβία η Πολωνική Προεδρία οργάνωσε μία συζήτηση στην οποία κάλεσε τους Υπουργούς Κοινωνικών Υποθέσεων στην Ευρώπη για να μιλήσουμε για τις καλές πρακτικές όσον αφορά στις μητρικές άδειε. Και βάσει τη συζήτηση στην Κρακοβία η Πολωνική Προεδρία συμμετείχε και την έκτακτη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είπε ότι το Συμβούλιο δεν θα δεχθεί 20 εβδομάδες μητρική άδεια με πλήρη, με πλήρη μισθό. Βέβαια βλέπουμε να υπάρχει το, να, να, να ανοίγει λίγο ορίζοντα και να υπάρχει και μια ευελιξία εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα. Και αυτό το αποδεικνύει και ένα ψήφισμα το οποίο θα παρουσιαστεί ή μάλλον καλύτερα παρουσιάστηκε την 1η Δεκεμβρίου. Το Συμβούλιο θέλει να συνεχίσει συνεργάζεται γύρω από αυτό το θέμα και θέλει να ευχαριστήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την τόσο καρποφόρα συνεδρίαση. το άνοιγμα του Συμβουλίου στις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο θα εξαρτηθεί και από την ευελιξία που θα επιδείξει το Κοινοβούλιο. Πολλά κράτη-μέλη μίλησαν για το θέμα της άρσης του συνταξιοδοτικού ορίου, της άρσης του ορίου Εμείς θέλουμε να έχουμε δημόσιες πολιτικές επικεντρωμένες γύρω από τον τομέα της εργασίας. Με δυνατό, με συνταξιοδότηση όσο το δυνατόν αργότερα. Διότι υπάρχει το θέμα της συνταξιοδοτικής ηλικίας, όπως προβλέπεται από τον νόμο, αλλά μετά έχουμε και το θέμα κατά πόσο απασχολείται ο ηλικιωμένος υπό το φως της χρηματοπιστωτικής κρίσης θα συνεχίσουμε με τη Δανέζικη Προεδρία να συζητάμε το θέμα. Και ελπίζουμε λοιπόν και από, και από τη Δανέζικη Προεδρία να κρατήσει αυτό το θέμα ως προτεραιότητα. Όσον αφορά τώρα στην απασχόληση των νέων και των ηλικιωμένων για να προσεγγίσουμε τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 δηλαδή να έχουμε το 75% απασχόληση μέχρι το 2020 θα χρειαστεί να αυξήσουμε την απασχόληση τόσο μεταξύ των νέων όσο και μεταξύ των ηλικιωμένων. Οι ηλικιωμένοι δεν κλέβουν τη δουλειά από τους νέους, όπως είπε και ο γερουσιαστής Αουγκουστίν. Δεν πρέπει να κηρυχθεί πόλεμος για τη δουλειά μεταξύ γέρων και νέων. Θα πρέπει αντί για πόλεμο εμείς να έχουμε ένα σύμφωνο υπέρ της απασχόλησης. Όπως είπε και κάποιος συνάδελφος πρέπει να δημιουργήσουμε πλήρη απασχόληση, συμφωνώ απόλυτα. Η εργασία για τους νέους συζητήθηκε ιδιαίτερα σε μια συνεδρίαση στο Συμβούλιο. Εμείς έχουμε ευθύνη έναντι των νέων, γι' αυτό λοιπόν εγώ υποστηρίζω ότι χρειάζεται μια ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, είναι θεμελιώδες αυτό. Εμείς πολύ συχνά μιλήσαμε για αυθεντική αλληλεγγύη, αλληλεγγύη με αλφα κεφαλαίο μεταξύ των γενεών, διότι η αλληλεγγύη δεν είναι μονόδρομος. Πρόκειται για ένα δρόμο διπλή, διπλής κατεύθυνσης. Θυμήσαμε και το θέμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Η κυρία Γιατσλοβιέτσκα μίλησε και είπε ότι θα πρέπει να παρακολουθήσουμε ποια είναι η αποτελεσματικότητα της χρήσης των κονδυλίων του ΚΤΕ. Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει και το σωστό συμπέρασμα της συζήτησής μας σήμερα. Και ανακεφαλαιώνοντας και κλείνοντας ευχαριστώ όλους τους βουλευτές, ευρωβουλευτές και εθνικούς βουλευτές για αυτή τη συζήτηση όπως είπε και ο συνάδελφος Ματίας Νουνιές από το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο οι πολιτικοί δεν πρέπει να σκέφτονται τις επόμενες εκλογές αλλά τις επόμενες γενιές. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω αυτά τα οποία έχω ήδη πει ή αυτά τα οποία ακούστηκαν. Το θέμα είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Είναι σαφές ότι δεν θα πρέπει να ολιγορήσουμε και θα πρέπει να πάρουμε μέτρα έτσι ώστε στα πλαίσια της στρατηγικής του 2020 να πετύχουμε τους στόχους μας. Η απασχόληση των νέων, τα θέματα της εσωτερικής μετανάστευσης που μπορεί να είναι ευεργετική για μία χώρα ή αρνητική και καταστροφική για άλλες χώρες. Το θέμα της εξωτερικής μετανάστευσης είναι κάτι το οποίο έχουμε βιώσει εδώ και δεκαετίες. Είναι δύσκολο να λυθούν όλα τα προβλήματα τα οποία θέτει. Είναι δύσκολο να καλύψουμε πλήρως και με σωστό τρόπο τις ανάγκες των μεταναστών τα θέματα της κοινωνικής συνοχής επίσης τίθενται ξεκάθαρα. Όλα αυτά τα προβλήματα βέβαια τα οποία τίθενται σήμερα δεν είναι πρόσφατα. Και ένα σχόλιο το οποίο θα ήθελα να κάνω σε τρία σημεία. Πρώτον, θα ήθελα να πω θέλουμε πράγματι εμείς να διατηρήσουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο τα επόμενα χρόνια. Σε ποιο βαθμό μπορούμε να κάνουμε αλλαγές, πρέπει να κάνουμε αλλαγές και σε ποιο βαθμό οι Ευρωπαίοι που έχουν δουλέψει για ένα τέτοιο πρότυπο θα πετύχουν να, το αλλάξουν. Χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχουν χώρες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν ισχυρά κοινωνικά συστήματα και ταυτόχρονα έχουν και χαμηλά ε, προϋπολογισμούς στον τομέα των κοινωνικών δαπανών. Λοιπόν, δεν θέλω να ονοματίσω τις χώρες αυτές, τις μεν και τις δε, αλλά τέτοιες χώρες υπάρχουν. Πρέπει λοιπόν εμείς να υπερασπιστούμε τα κοινωνικά μας πρότυπα με μεγαλύτερη ευθύνη και με σωστές ενέργειες. Αυτό είναι το μέλλον μας το οποίο σήμερα διακυβεύεται. Δύο άλλα θέματα τα οποία γίνονται όλο και περισσότερο σημαντικά σήμερα και τους δίνουμε νομίζω την απαιτούμενη σημασία, ιδιαίτερα σε μια εποχή δραματικής κρίσης. Από τη μία, η γύρανση της κοινωνίας. Είναι σαφές ότι πρέπει να δώσουμε σωστές απαντήσεις στα προβλήματα συνταξιοδότησης των εργαζομένων και των συνταξιούχων πώς μπορούμε να απασχολούμε αυτούς οι οποίοι μερικές φορές θέλουν και μπορούν να δουλέψουν μετά τα 50, μετά τα 60 και μετά τα 70, γιατί όχι. Εφόσον είναι υγιείς, γιατί να μην το κάνουν. Ευτυχώς το προσδόκιμο ζωής μας έχει ε, πράγματι αυξηθεί. Μπορούμε να πετύχουμε λοιπόν τους στόχους μας προωθώντας την απασχολησιμότητα των ε, ηλικιωμένων ε, πολιτών στην Ευρώπη. Πρέπει να προωθήσουμε λοιπόν τα πρόσωπα αυτά, πρέπει να προωθήσουμε τις ικανότητές τους σε επίπεδο εθνικό, σε επίπεδο περιφερειακό και τοπικό. Και παράλληλα έχουμε το θέμα της γεννητικότητας. Το θέμα της γεννητικότητας είναι δραματικό σήμερα για κάποιες περιοχές ήταν σοβαρό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να δώσουμε βοήθεια στις οικογένειες να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών και τις ανάγκες ε, της παρουσίας τους στον επαγγελματικό χώρο. Λοιπόν, αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία τέθηκαν, ακούστηκαν πολλές ιδέες, πρέπει να βοηθήσουμε έτσι ώστε να αλλάξουν κάποια πράγματα, Ακόμα και οι άνδρες γονείς, σαν παράδειγμα, θα πρέπει να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο από αυτόν που παίζουν σήμερα στην ανατροφή των παιδιών. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στην παρουσία του άνδρα και της γυναίκας στο σπίτι, στην οικογένεια, στα παιδιά πρέπει να προσέξουμε γιατί ε, πάρα πολλές γυναίκες, ένα μεγάλο ποσοστό των γυναικών αφιερώνουν την ενέργειά τους και το χρόνο τους στην ανατροφή των παιδιών και έτσι δυσκολεύονται να απασχοληθούν επαγγελματικά. Λοιπόν, βλέπουμε ποια είναι τα προβλήματα, βλέπουμε πώς τα προβλήματα οξύνονται από την εποχή της κρίσης στην οποία ζούμε, οι ερωτήσεις ε, τίθενται, κάποιες από αυτές θα συζητηθούν στις 8 και 9 Δεκεμβρίου στο Συμβούλιο, αλλά το θέμα το πρέπει να το αντιμετωπίσουμε νομίζω και μόνοι μας. Ελπίζω σε 2-3 χρόνια να μπορέσουμε να μπούμε σε μια νέα περίοδο ευημερία στην Ευρώπη και να αντιμετωπίσουμε τα δημογραφικά προβλήματα της Ευρώπης και το πρόβλημα της γύρανσης της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν αυτές τις μέρες συζητήθηκαν με ικανοποιητικό τρόπο και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας εδώ, να ευχαριστήσω και τα μέλη του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και είπατε ό,τι ήθελα να πω. Τα πήρατε από το στόμα μου. δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το δημογραφικό πρόβλημα, το ξέρουμε, το έχουμε μπροστά μας εδώ και καιρό και ξέρουμε ότι οι μεγάλες χώρες θα είναι αυτές που θα έχουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι Παράλληλα με την οικονομική πολιτική υπάρχει και η κοινωνική πολιτική. Όπως θέλουμε να λύσουμε τα οικονομικά προβλήματα, εξίσου θα πρέπει να λύσουμε και τα κοινωνικά προβλήματα. Διότι το ρίσκο είναι να παρέμβουμε αργά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιβιώσει αλλά θα πρέπει να λάβει υπόψη της το ρίσκο ότι αυτά τα δημογραφικά προβλήματα θα λυθούν ακόμη πιο δύσκολα στο μέλλον και θα πρέπει για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα να χρηματοδοτήσουμε ακόμη περισσότερα κονδύλια. Η Πολωνία περνάει αυτούς τους χαλεπούς καιρούς της κρίσης χωρίς να υπόκειται σημαντικές, σε σημαντικές ζημιές. Δεν είχαμε ποτέ αρνητική ανάπτυξη. Εντάξει, είμαστε πιο ήσυχοι στην Πολωνία σχετικά. Αλλά οι ελίτ ανησυχούν το ίδιο. Και εμείς θα πρέπει να ετοιμαστούμε. Ξέρω ότι ο πρόεδρος της Γερουσίας και ο πρόεδρος του ΣΕΜ έχουν την υποχρέωση να κλείσουν αυτή τη συνάντηση. τον πρόεδρο του Πολωνικού ΣΑΕΜ να μας κλείσει. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε πρόεδρε της Γερουσίας, πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αντοχή σας, για την ενεργή σας συμμετοχή σε αυτήν τη συζήτηση για θέματα τόσο σημαντικά. Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες. όλους όσους θέλησαν να ονομάσουν τα προβλήματα, λέγοντας ότι είναι προβλήματα που αφορούν σε όλους μας, σε όλους μας τους πολίτες. Ευχαριστώ. Πέρας της συνεδρίας.